Cari colleghi, diamo inizio ai nostri lavori. Ξεκινάμε συνάδελφοι με κάποια μικρή καθυστέρηση. Αλλά ακόμα και τώρα, παρότι περιμέναμε 15 λεπτά, δεν έχουν έρθει πάρα πολλοί συνάδελφοι, αλλά δεν θα καθυστερήσουμε άλλο. Πρώτο θέμα, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση του Κωσυφοπεδίου. Η η συνάδελφος Λούνατσεκ. Πριν της δώσω το λόγο θα ήθελα να σας ενημερώσω αν δεν το ξέρετε ότι αύριο στις 6 το απόγευμα θα υπάρξει μια έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής μας με τον Πρωθυπουργό του Κοσφοπεδίου και με τον Υπουργό και τον Υπουργό εσωτερικών υποθέσεων και τοπικών αρχών Πέτροβιτς, Σλόμπονταν Πέτροβιτς. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφου που ήρθαν εδώ για να παρακολουθήσουμε την πρώτη εκδοχή της έκθεσής μου για το Πέδιο. Συζητούμε για όλες τις χώρες διεύρυνσης μετά από την έκδοση της έκθεσης των εκθέσεων πρόοδου από την Κομισιόν και θα ήθελα να διεξέλθω μερικά από τα κύρια θέματα τα οποία είναι για μένα σημαντικά και προσβλέπω σε περαιτέρω συζήτηση με τους συναδέλφους. Γνωρίζοντας ότι το θέμα αυτό είναι αμφίμαχο για ορισμένα θέματα, για ορισμένα σημεία, ελπίζω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ευρία πλειοψηφία στις κύριες πτυχές του. Στην έκθεση αυτή, καταρχήν, μπορώ να επιβεβαιώσω και θέλω να το πράξω ότι η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει για το κοσφοπέδιο. Πρέπει να συνεχίσει δηλαδή η διαδικασία διεύρυνσης και επίσης και το ευρωπαϊκό εγχείρημα ειρήνευσης δεν θα μπορέσει να ευδοκιμήσει πλήρως εάν δεν έλθουν όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων εν καιρό και ελπίζω σύντομα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε και πάλι αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών αυτών και πρέπει να το πράξουμε και για το ίδιο το Κωσυφοπέδιο. Όπως και στην τελευταία μου έκθεση, θα ήθελα να χαιρετήσω τα τελευταία, να, να καλέσω μάλλον τα τελευταία πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν αναγνωρίσει το Κωσυφοπέδιο να το πράξουν. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία ομοφωνία για τα θέματα αυτά στο Κοινοβούλιο. αλλά ξέρουμε ότι η πλειοψηφία συμφωνεί για το θέμα αυτό. Επίσης θέλω να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη τονίσει και στο παρελθόν και έχει ανανεώσει η διεθνή κοινότητα την εστίασή της στο Κωσυφοπαίδιο, ιδίως μετά τις δηλώσεις κάποιων Σέρβων πολιτικών που ζήτησαν τη διχοτόμηση του Κωσυφοποδίου κοσφοπεδίου. Αυτό το απορρίπτω διαρρήδιν όπως έχει πράξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή τη δυνατότητα διχοτόμησης του κοσφοπεδίου. Στην ομάδα εργασία για τα Δυτικά Βαλκάνια είχαμε συναντηθεί με εκπροσώπους του Κοινοβουλίου του Κωσυφοπέδιου και νομίζω ότι κάποιοι εκπρόσωποι είναι παρόντες εδώ, θα ήθελα να τους καλωσορίσω αυτοί που είναι εδώ από το Κωσυφοπέδιο και είχαμε τονίσει ότι και ο διάλογος για τις υποξενικές θεωρήσεις, τις βίζες, είναι ουσιώδης για τους πολίτες του Κοσμοπεδίου ανεξάρτητα από την εθνοτική τους προέλευση. Είτε είναι ε, Αλβανοί, Σέρβοι, Ασκάλοι, Αιγύπτιοι, Ρώμα κτλ. Ελπίζω λοιπόν ελπίζω ότι η διατύπωση στην έκθεση του κυρίου Φιούλε που λέει ότι πρέπει εφέτος να ξεκινήσει ο διάλογος για τις προξενικές θεωρήσεις, ότι θα υλοποιηθεί και θα ξεκινήσει η Κομισιόν το διάλογο έχοντας ήδη ένα οδικό χάρτη. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση του Κωσόβου μπορεί να κάνει όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσει τη φιλελευθερωποίηση παροχής βίζας για τους πολίτες της. Η κατάσταση τώρα στο ίδιο το Κώσοβο. Στην έκθεση εκφράζω τη λύπη μου για τις σοβαρές ατασταλίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, το μακρό διάστημα που χρειάστηκε για να υπάρξει ένα κοινοβούλιο και εκλογή του Προέδρου του και επίσης σχηματισμός κυβέρνησης. Επίσης αναφέρθηκα στην ανάγκη να υπάρξει ταχύτης σε ό,τι αφορά την τιμωρία των υπετίων για, την, για τις απάτες και την οθεία κατά τη διάρκεια των εκλογών και την ανάγκη να σταματήσει η κουλτούρα τιμωρησίας που σοβεί σε, πολλά, σε πολλές περιπτώσεις στο κοσμοπέδιο, ότι πρέπει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Έρχομαι τώρα σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο διάλογος μεταξύ Σερβίας και κοσφοπεδίου. ευτυχώς επαναλήφθηκε φέτος και είδαμε και μια ανακοίνωση τύπου όπου αναφέρεται ότι υπήρξε θετική επανέκτηση επανέναρξη του διαλόγου. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος συνεργασίας και μελλοντική συνεργασία μεταξύ της Σερβίας και του Κωσυφοπεδίου. Ελπίζω ότι ο διάλογος αυτός θα έχει θετική απόλυξη, ότι οι συμφωνίες οι οποίες έχουν ήδη επιτευχθεί θα υλοποιηθούν και από την σερβική κυβέρνηση το ταχύτερο δυνατό. Και αναφέρθηκα στο θέμα αυτό με την ελπίδα ότι με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί το έδαφος για μια συμφωνία σε επίσημο επίπεδο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κωσυφοπεδίου. Η τεταμένη τώρα και ασταθής κατάσταση στο βορρά του Κωσυφοπεδίου είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ανησυχίε σε όλους την περιοχή και φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσκαλώ και πάλι την κυβέρνηση της Σερβίας να, διαλύσει τις παράλληλες δομές και να δώσει μια ευκαιρία στο σχέδιο Αχτισάρι και στο Βορρά. Θα ήταν πολύ θετικό να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο. Οι Σέρβοι αυτοί οι οποίοι δέχονται στο βόρειο μέρος του Κωσυφοπεδίου να μείνουν εκεί θα μπορούν να έχουν ένα ευρύ πεδίο αυτονομίας, εάν το επιθυμούν. Και επίσης στο νότιο τμήμα του Κωσυφοπεδίου, στο ΙΜΠΑ, υπήρξε σημαντική πρόοδος, έχουν εκλεγεί τοπικοί άρχοντες ε, δήμαρχοι, κοινοτάρχες, υπήρξε μια πρόοδος και στα οικονομικά θέματα στις κοινότητες αυτές. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά για να εξασφαλιστεί ο πολυεθνικός χαρακτήρας του κοσυφοπεδίου εν γέννη. Το κράτος δικαίου και η σημασία του κράτους δικαίου είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλοι. Η Eurolex, η Eurolex είναι η μεγαλύτερη δύναμη που έχουμε στην Ευρώπη ως Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει σημαντικό ρόλο σε όλο το τομέα της καταπολέμησης διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Ο κ. Λιμάη, ο πρώην Υπουργό Μεταφορών αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέταση και μπορεί να παραπευθεί σε δίκη. Υπάρχουν λοιπόν ενέργειε κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Εκεί η κυβέρνηση του Κωσικοπέδου πρέπει να πράξει περισσότερο. Αυτό το οποίο ζητώ από την πλευρά των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτών των χωρών που έχουν τμήματα στην ULEX είναι να δείξουν μεγαλύτερη ευελιξία στο να αποσπάσουν δικαστές και ανακριτές στη ULEX γιατί χρειάζονται και επίσης να βοηθήσουν να υλοποιηθεί το πρόγραμμα προστασίας ε, μαρτύρων στο Κόσοβο και να δεχτούν ότι κάποιοι από αυτούς θα πρέπει να μετακινηθούν σε, άλλα, σε άλλους τόπους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί πρέπει να βοηθήσει η σύνολη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκα λοιπόν και στα μέλη της συνέλευσης του Κωσικοπαιδίου που είναι παρόντες. Η συνέλευση αυτή έχει να διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να ελέγξει την κυβέρνηση σε θέματα προπολογισμού σε σχέση με τη διαδικασία μεταρρύθμισης του εκλογικού κώδικα και επίσης παροτρύνω την ε, συνέλευση του Κωσικοπαιδίου να προχωρήσει σε αυτές τις υπεσχημένες στην κοινή γνώμη μεταρρυθμίσει. μεταρρυθμίσεις μέσα στα πλαίσια των 18-24 μηνών που ακολουθούν τι εκλογέ και όχι να τι παραπέμψει σε ελληνικέ καλένδε. Ανεφέρθηκα στη διαφθορά, εξακολουθεί να είναι κάτι το οποίο απασχολεί πολύ του πολίτε του πεδίου και η κυβέρνηση πρέπει εκεί να πράξει πολλά και επίσης και οι ιδιοκτικέ αρχές και οι αστυνομικέ αρχές θα πρέπει να πράξουν τα απαραίτητα ώστε να καταλάβουν οι πολίτες ότι θα σταματήσει αυτή η διαφθορά και να μπορέσουν να επανακτήσουν εμπιστοσύνη στο κράτο δικαίου για τη δικαστική εξουσία. Υπήρξε κάποια πρόοδο στη μεταρρύθμισή της, αλλά ακόμα η ανεξαρτησία των δικαστών από την πολιτική εξουσία και ο επαγγελματισμός τους είναι το μίσο που χρειάζεται ακόμα περαιτέρω προσπάθειες. Επίσης και ο δημόσιος μηχανισμός, οι δημοσίοι υπάλληλοι, για μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απαραίτητο να είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες και υπόλογοι για να λειτουργήσουν σωστά οι κρατικοί θεσμοί είναι πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ίδιο του στο κράτος. Ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μονάχα στο Κωσυφοπέδιο και τα Βαλκάνια, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εκεί η ανάγκη να έχουμε ισχυρά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι κεφαλαιώδης. Οι διακρίσεις σε εθνοτικό επίπεδο, σε επίπεδο ηλικίας, ε, σεξουαλικού προσανατολισμού, λόγω ηλικίας κτλ. Όλα αυτά εξακολουθούν να είναι προβλήματα στη χώρα αυτή. Υπάρχει καλό νομοθετικό επίπεδο, αλλά δεν υπάρχει επαρκή εφαρμογή της νομοθεσίας. Χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη η εφαρμογή του νόμου. Θα ήθελα να ζητήσω να υπάρξει και περισσότερη υποστήριξη στο έργο του Διοικητικού Επιτρόπου. Πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά. Και εκεί υπήρξε κάποιο πρόοδο αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει νέα νομοθεσία, ιδίως για το ιστορικό κέντρο του Πρίζρεν, το οποίο θα πρέπει να προστατευτεί, να τύχει προστασίες και υπάρχουν κάποια νομικά στοιχεία που ελείπουν αυτή τη στιγμή από, την, από το συνολικό πλαίσιο. Υποστήριξη κοινωνίας των πολιτών, αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων, η κατάσταση του περιβάλλοντος, όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα. Ξέρω τα προβλήματα των δύο ε, θερμικών σταθμών ενέργειας του Κόσοβο Α και Κόσοβο Β που και άνθρακα και δημιουργούν πολλά προβλήματα στους ε, πολίτες και κυρίως στα παιδιά που ζουν στην περιοχή της Πριστίνα όταν γεμίζει από εθάλιο αέρας από την καύση άθρακος από τους σταθμούς Α και Β. Είναι απαραίτητο να υπάρξει περισσότερη επένδυση σε ανανεώσιμες ενέργειες, σε αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και επίσης να βρούμε έναν τρόπο να υπάρξει μια ε, μελέτη για ένα τρίτο θερμικό σταθμό καύσεως άνθρακα στο Κοσμοπέδιο και να κλείσει τουλάχιστον ο σταθμός Κόσοβο 1 το ταχύτερο δυνατό. Αυτά είναι τα κυριότερα λοιπόν θέματα τα οποία εγώ ήθελα να σας αναφέρω. Η ελπίδα μου είναι ότι μαζί με τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή συζήτηση. Ξέρω ότι παραμένουν κάποιε διαφορέ μεταξύ μα σε σχέση με το καθεστώ Κωσυφοπέδιου κτλ. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε την ευρεία πλειοψηφία που έχουμε επιτύχει και να εξασφαλίσουμε ότι το Κόσοβο θα έχει ένα μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήμασταν αυτοί που υποστήριξαν περισσότερο τη διαδικασία αυτή στο κοσυφοπαίδιο και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συζήτηση ακόμα και αν δεν συμφωνήσουμε όλοι και τελικά θα καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση η οποία θα ψηφιστεί στην Ορομέλεια τον επόμενο Μάρτιο και προσβλέπω στα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Προηγουμένως αναφερθήκατε στην παρουσία μιας αντιπροσωπείας από την κοινοβουλευτική ε, συνέλευση του Κοσμοπεδίου δεν ήταν παρόντες τότε, αλλά τώρα φτάνουν και επομένως τους χαιρετούμε και τους ευχαριστούμε στην, για την παρουσία τους. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Κούκαν, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της αντίστοιχης αντιπροσωπείας και για το κοσφοπέδιο. Σας παρακαλώ αν μπορείτε να παραμείνετε μέσα σε τρία λεπτά. Δεν θέλω να είμαι άκαμπτος, αλλά προσπαθούμε να οργανώσουμε με τον καλύτερο τρόπο το χρόνο μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την έκθεση της κυρίας Λούνατς και είναι καλή βάση για το Κοινοβούλιο την εισήγηση για το κοσυφοπαίδιο. Είναι η συνήθις φράση πρωτού αρχίζει κανείς την παρουσίασή του, αλλά εγώ το πιστεύω διότι νομίζω ότι το κείμενο αναφέρει όλα τα πιεστικά θέματα και ελπίζω ότι η εισήγηση θα βοηθήσει το κοσυφοπαίδιο να προοδεύσει στις ε, μεταρρυθμίσεις και σε όλο το πρόγραμμα ολοκλήρωσης. Διότι πιστεύουμε όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του κοσυφοπεδίου ε, μέχρι τώρα, ότι όλοι βλέπουμε το μέλλον του κοσυφοπεδίου στην Ευρώπη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με την αξιολόγηση της Επιτροπής που εκφράστηκε στην έκθεση προόδου ε, το Κωσυφοπαίδιο έχει κάνει πρόοδους σε πάρα πολλούς τομείς πολιτικής, κυρίως ε, στο συντονισμό του ε, Ευρωπαϊκού Προγράμματος το Κωσυφοπαίδιο έχει προοδεύσει και μερικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως στον δικαστικό τομέα, εξακολουθούν να υλοποιούνται. Το, ο διάλογος με το Βελιγράδι έχει ξεκινήσει και πάλι και ελπίζω ότι θα αποφέρει απτά αποτελέσματα τόσο για τη Σερβία όσο και για το Κωσυφοπέδιο. Ίσως να είμαι πολύ αισιόδοξο παρόλο που γνωρίζω τις δυσκολίες, αλλά είναι καλό να είναι κανείς αισιόδοξο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι όλη η διαδικασία ξεκίνησε ούτως ώστε η ζωή των πολιτών του Κωσυφοπεδίου και της Σερβίας να διευκολυνθεί παρόλο που πολλές εξελίξεις στο τελευταίο εξάμεινο δείχνει ότι καμιά φορά το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο. Θα έπρεπε λοιπόν ενεργά να υποστηρίξουμε και τις δύο πλευρές τις προσπάθειές τους να εργαστούν για τα θέματα του διαλόγου. Είναι επίσης σημαντικό να επισημάνουμε ορισμένα προβληματικά θέματα. Το κοσυφοπαίδιο θα πρέπει να επιτυχιαχύνει τις ικανότητες δημόσιας διοίκησης, επιβολής νόμου και θα πρέπει οι δικαστικές αρχές να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα. Δεν είναι μόνο η ειδικότητα του κοσφοπεδίου βέβαια στο οργανωμένο έγκλημα. Η κατάσταση στο Βορρά είναι ακόμη ε, πάρα γεμάτη ένταση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε διάφορες ομάδες να αποφασίζουν τις εξελίξεις σε αυτό το τμήμα του κοσφοπεδίου. Ενώ δεν έχουμε καμία αντίρρηση στα δικαιώματα των πολιτών για διαδηλώσεις ειρηνικές, θα πρέπει η Ιούλεξ και η ΚΕΙΦΟΡ να ασχοληθούν. Η Ιούλεξ αναφέρθηκε από την κυρία Λούνατσεκ και νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την αποστολή της δύναμης αυτής στο Κωσυφοπαίδιο, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και τη σημασία της αποστολής αυτής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν καλή ιδέα να έχουμε μια συνάντηση με εκπροσώπους της Ιούλεξα και να έχουμε από πρώτο χέρι επικαιροποίηση της κατάστασης εκεί. Σχετικά με την απελευθέρωση των θεωρήσεων, χαίρομαι που η Κομισιό ε, πρότεινε να, την έναρξη διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό. Δεν πρέπει να αφήσουμε πίσω το κοσυφοπαίδιο και να απομονώσουμε τους πολίτες από την υπόλοιπη Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές του κοσυφοπαιδίου θα πρέπει να επιδείξουν σαφή πρόοδο και αποφασιστικότητα εργαζόμενες για να εκπληρωθούν οι όροι που απαιτούνται για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεωρήσεως. Ελπίζω να έχουμε καλή συνεργασία για αυτή την εισήγηση. Η προθυμία του εισηγητού αναγνωρίζεται και εμείς θα αντιδράσουμε κατά συνέπεια. Ευχαριστώ. κύριε Κούκαν. Ο κύριος Πανσέρη έχει τον λόγο, σκιώδης, ως εισηγητής για τη σοσιαλιστική ομάδα. Τρία λεπτά, αν μπορείτε, παρακαλώ. Βεβαίως. Γιατί βρισκόμαστε και σε επίπεδο πρώτης συζήτησης, θα υπάρξει η ευκαιρία να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι η πρόταση οδηγη... Ε, εκθέσεως έχει ορισμένα στοιχεία τα οποία επικροτώ. Καταρχήν την προοπτική για ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βέβαια αυτό πρέπει να γίνει παράλληλα με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την Σερβία, γιατί πιστεύω πρέπει να υπάρξει παραλληλισμός για τις δύο αυτές χώρες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα και που όπως αναφέρθηκε αφορούν το κράτος δικαίου που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι το κοσυφοπέδιο θα είναι σε θέση να έχει οικονομική ανάπτυξη, να είναι αξιόπιστο σε ευρύτερο επίπεδο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τα κονδύλια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που τελικά μπλοκαρίστηκαν λόγω ανητικών στοιχείων που ανέκυψαν μετά από την παρακολούθησή τους που οφείλονται σε ορισμένε αποφάσεις του, της κυβέρνησης, συγκεκριμένα την πώληση της τηλεφωνικής εταιρείας του Κωσικοπαιδίου. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό και πάνω απ' όλα υπάρχει, και θέλω να σταθώ λιγάκι στο θέμα αυτό, κάτι για την EULEX, την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω την ίδια ενθουσιώδη άποψη όπως η κυρία Λούνατσερ για την αποστολή αυτή, ιδίω σε σχέση με την αναχρηματοδότηση που προβλέπεται για τον Ιούλιο του 2012. Νομίζω ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε πολλά σημεία σε ορισμένε περιπτώσει δεν υπήρξε η, απολ, η απαραίτητη λειτουργία και απόδοση της ε, ε και υπήρξε και μια έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της EULEX η οποία επηρέασε και τον επαγγελματικό της χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητά της επιτόπου. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα όπως αυτό. Εάν παραμείνει με αυτή τη μορφή η Ιούλεξ, θα πρέπει να υπάρξει μια σειρά μεταρρυθμίσεων και ελέγχων και το λέω στεναρά ότι θα πρέπει και η έκθεση να αναφέρει και κάποια από τα σημεία στα οποία είναι απαραίτητο να υπάρξει μια διόρθωση πορείας σε σχέση με την EULAX στο κοσφοπέδιο. Γιατί αν θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθεί αυτό που ζητάει η κυρία Λούνετσεκ σε σχέση με τη μελλοντική πορεία της χώρας αυτής, τότε θα πρέπει να παρέμβουμε με μεγαλύτερη γαλήνη και με μεγαλύτερη σοβαρότητα μέσω της, με της αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνω εδώ, αλλά θα επανέλθω εάν χρειαστεί σε περαιτέρω συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν ακριβώς τα τρία λεπτά. Μπράβο. Ο κύριος Σαλάκη, αν, μπορείτε και εσείς τα τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ δεν είμαι και τόσο ενθουσιώδης σχετικά με τον γενικό τόνο της έκθεσης, την έλλειψη κριτικής ε, σχετικά με την κατάσταση στο κοσυφοπαίδιο. Δεν είναι καλή ε, συνεισφορά στην ε, μεταρρύθμιση των θεσμών του κοσυφοπαιδίου και νομίζω ότι η έκθεση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση στο κοσυφοπαίδιο που δεν είναι τόσο ρόδινη όπως εμφανίζεται εδώ. Υπάρχει πάντοτε το μεγάλο ανοιχτό θέμα πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν αγνωρίσει αυτή την οντότητα και έχουν καλούς λόγους που δεν την αναγνωρίζουν. Δεν βλέπω και τόσο μεγάλη ε, πρόοδο κατά την κρίση πολλών διεθνών οργανισμών σχετικά με την πρόοδο στο κοσυφοπαίδιο στο δρόμο του κράτους δικαίου και της ολοκλήρωσης ε, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Νομίζω ότι η αξιολόγηση είναι γενικά αρνητική και συμφωνώ. Δεν είδα καμία σημαντική προσπάθεια. Αν θέλουμε να κρίνουμε τα γεγονότα, και όχι με, τα συνήθη, με τις συνήθεις λέξεις και τη συνήθη γλώσσα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο κοσυφοπέδιο, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το κρίσιμο θέμα της Ιούλεξ. Οι εκπρόσωποι της Ιούλεξ και οι πολιτικοί θύνοντες ήρθαν εδώ πριν μερικούς μήνες και, και τα γεγονότα ε, που παρουσίασαν δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά. Η Ulex είναι ένα περίεργο όργανο που θα πρέπει να είναι σύμβουλη στην κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου, ενώ ε, στην πραγματικότητα θα έπρεπε να αντικαταστήσουν ε, το δικαστικό σώμα, το γραφείο του ισαγγελέα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος κοστίζουν 1,5 ε, εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στους φορολογούμενους. Είναι λοιπόν τρομερό το ποσό αυτό για λιγότερο από 200 άτομα, 2.000 άτομα. 100 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό με συγχωρείτε και δεν ε, ξέρουμε τα αποτελέσματα. Αυτά αποτελέσματα διάβασα την έκθεσή τους ε, και υπήρχε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την έκθεση, η οποία είναι κατανόητη. Δεν μιλάνε για τίποτα σημαντικό που να έχουν πραγματοποιήσει στον τομέα αυτό. Πώς χρησιμοποίησαν τα χιλιάδες άτομα αυτό το προσωπικό ε, και όλα τα χρήματα τα ευρωπαϊκά. Είναι αδύνατο να το κατανοήσει κανείς από την έκθεση του ρώτησα και η απάντησή τους δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική. Νομίζω ότι η έκθεση ε, θα έπρεπε να κατακρίνει πολύ περισσότερο την ε, απόδοση της Ιούλεξ και θα ήθελα να πω στην Αλφα Παντζέρη ότι θα πρέπει ε, και πάλι να ξαναδούμε τι γίνεται με αυτό το όργανο και να αλλάξουμε την οργάνωση και να του ζητήσουμε να είναι πιο αποτελεσματική και πρώτα απ' όλα να είναι αξιόπιστοι σε αυτά που κάνουν. Ευχαριστώ κύριε Αρλάκη. Ο Earl of Dartmouth έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τη στιγμή που ήρθα στην αίθουσα αυτή έχω σημειώσει κάποιες από τις λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με το κοσυφοπαίδιο. Διακρίσεις. Δικαστική εξουσία. Αρνητική λειτουργία του κράτους δικαίου. Διαφθορά έλλειψη ελεύθερου τύπου. Ε, οργανωμένο έγκλημα. Ξέπλυμα χρημάτων. Αυτή ήταν, αυτή ήταν η όρη που χρησιμοποίησαν οι συνάδελφοι για να περιγράψουν την κατάσταση στο Κωσφοπέδιο. Ίσως θα πρέπει να προσθέσουν και το λέει και η έκθεση ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η ανεργία επισήμω είναι 45% στο Κωσφοπέδιο. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία και σίγουρα θα είναι περισσότερο στην πράξη. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα δυσλειτουργικό κράτος, μια δυσλειτουργική κοινωνία. Μόνο μια ομάδα με τις αυτοκρατορικές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή η οποία είναι ικανοποιημένη με αυτή την κατάσταση της χώρας αυτής. Κανείς δεν θα μπορούσε να δεχτεί μια τέτοια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόμμα μου λοιπόν θα καταψηφίσει αυτή την κατεύθυνση, γιατί το κόστος αυτής της δυσλειτουργικής κοινωνία θα πρέπει να το επομιστεί πλήρω ο φορολογούμενος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχα καταθέσει μια σειρά από ερωτήσει προς την Κομισιόν πριν από δύο εβδομάδε περίπου και περιμένω αδειμόνω για την απάντηση για το πόσο υπολογίζει η Κομισιόν θα είναι το κόστος του κοσφοπεδίου. Αλλά η χώρα αυτή έχει πάρει ήδη 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια τα τελευταία 10 χρόνια η Σερβία και το 25 θα είναι κάτι το αντίστοιχο. Όταν αγωνίζονται να πληρώσουν τους βασικούς λογαριασμούς τους οι συμπολίτες μου, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ να δεχτούμε άλλο ένα κράτος το οποίο <clears throat> θα πρέπει να το ταΐζουμε. Γιατί κάτι τέτοιο είναι αυτό. Βλέπω επίσης ότι υπάρχει μια πρόταση, δεν ξέρω αν είναι σοβαρή αυτή η πρόταση, να υπάρξει φιλελευθερωποίηση προξενικών θεωρήσεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κωσφοπεδίου. Μα πώς μπορεί να γίνει αυτό μια αξιόπιστη πρόταση με το επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος το οποίο περιέγραψαν πάρα πολλοί συνάδελφοι στο Κωσφοπέδιο. Μια τελευταία παρατήρηση. Κάποια κόμματα στην Μεγάλη Βρετανία τον θεωρούν ότι είναι υπέρ ενός περιορισμένου προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω εκπροσώπους τους εδώ. <clears throat> Θέλω να τους πω, δεν είναι αξιόπιστη η θέση τους όταν λένε ότι θέλουν μείωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συγχρόνως θέλετε τη διεύρυνση με το Κόσοβο και άλλες χώρες της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ντάρτμουθ γιατί σεβάστηκε το χρόνο που είχε στη διάθεσή του. Βάιγκελ, τρία λεπτά. Η κατάσταση στο Κωσίφο πεδίο δεν είναι η καλύτερη δυνατή και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, είναι σαφές. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το Κωσυφοπέδιο με τόσο θα έλεγα βίαιη και καταστροφική ρητορική σαν και αυτήν την οποία ακούσαμε. Πρόκειται για μια νέα χώρα, περίπλοκη νέα χώρα, περίπλοκο νέο έθνος, λέει ο μιλητής. Και πολλά από τα προβλήματα του κοσυφοπεδίου προέρχονται από το ότι Επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τον έχουν ακόμα, δεν το έχουν ακόμα αναγνωρίσει. The fact is uh, that uh, it is difficult to build up. Είναι δύσκολο βέβαια να δημιουργήσει κανείς μια νέα χώρα, μια νέα κοινωνία και να αποκτήσει σχέσεις με τις υπόλοιπες χώρες, ιδιαίτερα τις γειτονικές χώρες. και μάλιστα όταν δεν υπάρχουν ομόφωνες απόψεις σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας αυτής. Πάντως νομίζω ότι εξ αυτού μπορεί κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα, στα συμπεράσματα μάλλον, με τα οποία προσπαθεί να εξηγήσει κανείς τις συγκρούσεις στα σύνορα ε, με τις γειτονικές χώρες. Αυτό έχει σημασία για τη σταθερότητα της Ευρώπης, τη σταθεροποίηση αυτής της περιοχής της Ευρώπης ε, και θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιεί μία γλώσσα απέναντί της. Είναι πραγματικά πολύ ευθυνό το να μπορεί να σπρώξει το κοσφοπέδιο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να πληρώσει το κόστος μιας μελλοντικής πολεμικής σύραξης. Συνεπώς συγχαίρω τον εισηγητή, την εισηγήτρια για την εξαιρετική της έκθεση. Την έχει συγγράψει καλή την πίστη και προσπαθεί να δώσει κίνητρα. Θα ζητήσω από την κυβέρνηση του Κοσφοπεδίου να είναι πιο δεκτική εν περιπτώσει απέναντι στους Σέρβους, να μπορέσουν να επιστρέψουν στο Κοσφοπέδιο και αυτοί οι Σέρβοι και να δώσει επίσης και μεγαλύτερο βάρος στο θέμα της προστασίας των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στη χώρα. Ευχαριστώ κύριε Βάιγκελ. Ο κύριος Τάνοκ, τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, διάβασα την έκθεση αυτή. Έχω βέβαια διαφορές απόψεων με την κυρία Λούνετσικ όπως και στο παρελθόν, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε γαλήνια γλώσσα όταν περιγράφουμε την κατάσταση του Κωσυφοπέδιου. Το Κωσυφοπέδιο όπως παραμένει ένα ανεπίλητο πρόβλημα για τη διεθνή κοινότητα και όχι μοναχά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μονάχα υπάρχουν πέντε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν το αναγνωρίζουν, αλλά έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το σύνολο του πλανήτη μας. Τουλάχιστον το μισό από τη Γενική Συνέλευση του, των Ηνωμένων Εθνών και δύο μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία, η Ρωσία και η Κίνα, δεν συμφωνούν με την αναγνώριση του κοσμοπεδίου. Αυτή είναι μια κατάσταση λοιπόν πολύ δύσκολη να είναι μια χώρα σε κατάσταση λίμπο που δεν μπορεί να είναι διατηρήσιμη στο δίνεκε. Το κοσμοπέδιο δυστυχώ χρειάζεται δυστυχώς πάρα πολλού διεθνεί φορεί να είναι παρόντε για να το βοηθήσουν ο ΣΑΙ και η ΦΟΡ, η ULEX και όλοι αυτοί κοστίζουν της Παναγιάς στα μάτια στους διεθνείς φορολογούμενους. Πάρα πολλά λεφτά για μια μικρή χώρα που δεν έχει έξοδο στη θάλασσα και μέχρι ότου υπάρξει σαφήνεια για το νομικό καθεστώς της χώρας αυτής θα υπάρχει και πρόβλημα με έλλειψη διεθνούς ε, άμεσης επένδυσης. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρά προβλήματα για να το πω επίοικος. Δυστυχώς το κοσφοπέδιο γίνεται όλο και περισσότερο μια μονοκουλτούρα, μια μονοκαλλιέργεια η υποστήριξη προς το Κοσφοπέδιο την εποχή του πολέμου με τη Ιουκοσλαβία είχαν σαν στόχο να μπορέσει να μείνει πολυπολιτισμικό μέρος το Κοσφοπέδιο. Αλλά αντίθετα βλέπουμε ότι φεύγουν όλο και περισσότερο οι Σέρβοι από το Κοσφοπέδιο. Πολλοί έχουν πάει στο βορρά, στην Μητρόβιτσα, που είναι μια περιοχή που είναι τώρα πια σχεδόν τελείως σερβική. Κάτω από τον, νότια από τον ε, ποταμό Ιμπάρ είναι σχεδόν μόνο αλβανικό το κοσφοπέδιο. Δεν ε, μπορώ να εκπροσωπώ, να όλη μου την ομάδα μου, αλλά εγώ έχω τονίσει πάντα ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια συζήτηση για τα θέματα αυτά και οι προσπάθειες κάθε Άστον και του Ρόμπερ Κούπερ πρέπει να στραφούν στο να βρεθεί μια ε, ανταλλαγή γης για ειρήνη, ώστε να μπορέσει να εξασφαλιστεί ένα αναγνωρισμένο διεθνές σύνορο του κοσμοπεδίου που να αναγνωρίζεται από τη Σερβία και τον υπόλοιπο κόσμο. Αν δεν θεωρεί η Σερβία ότι έχει καταλήξει σε μια θετική λύση με το να έχει την κυριαρχία στην περιοχή βόρεια από τον ποταμό Ήμπαρ ως ε, αντάλλαγμα για τους θυλάκους στο νότο και ίσως δίνοντας ένα τμήμα της περιοχής της κοιλάδας του Κωσόβου στους ε, που είναι αλβανοκρατούμενοι στο Κωσυφοπέδιο δεν θα πρόκειται να υπάρξει καμία λύση. Ζητάμε από τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς να έχουν μια λύση δύο κρατών. Γιατί λέμε λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει στην περίπτωση της Ευρώπης σε μια περιοχή που έχει εξίσου έντονες αντιμαχίες και μίση και δυσκολίες. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ανοιχτό μυαλό και να δούμε το θέμα μιας ανταλλαγής γης για ειρήνης, ώστε να υπάρξει συμφωνία και των υπολείπων μελών του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εξασφαλίσουμε ότι το Κωσυφοπέδιο θα έχει ένα ελεύθερο και θετικό μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Κύριε Σπρέντα, όχι πάνω από τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, για τα τρία λεπτά ε, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για την πρώτη παράγραφο. Νομίζω ότι είναι κάπως αφελής, διότι με συγχωρείτε που είμαι τόσο αυστηρός, αλλά νομίζω ότι τα πέντε χώρες που δεν αναγνωρίζουν ε, το κοσφοπέδιο είναι σημαντικό. Δεν είναι περιφερειακό ε, θέμα που, δε, που έχει ίσονα σημασία. Πρόκειται για ένα θέμα πολιτικό εξαιρετικά λεπτό. Και βρίσκω ότι η έκθεση δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτός. Είναι σαν η πλειονότητα των 22 χωρών που αναγνωρίζουν το κοσυφοπέδιο είναι ε, κάτι το αποδεκτό. Για τα πέντε άλλα είναι ένα λεπτό θέμα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πέντε αυτές χώρες σοβαρά και όχι να τις ε, παραβλέπουμε έτσι σε αυτή την παράγραφο που τις ε, καλεί να αναγνωρίσουν το κοσυφοπέδιο. Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι πριν από μερικές μέρες στον τύπο είδαμε μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία 20.000 Σέρβοι που ζουν στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο είχαν ζητήσει μια υποστήριξη για την προστασία τους στις ρωσικές αρχές και σύμφωνα με μερικά ε, σχόλια, ένας ικανός αριθμός Σέρβων στο Κωσυφοπέδιο θέλουν να αποκτήσουν ρωσική υπηκότητα. Μπορεί κανείς να ερμηνεύσει διαφορετικά, με διάφορους τρόπους αυτή την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι ενέχει σημασία. Γιατί δεν σκέφτονται εμά τους Ευρωπαίους. Αυτό δείχνει την έλλειψη εμπιστοσύνης που ένα μέρος του πληθυσμού του Κωσυφοπεδίου ε, ε, που δεν, δεν έχει εμπιστοσύνη και στις 22 χώρες που έχουν αναγνωρίσει το κοσμοπέδιο και στις 5 που δεν το έχουν αναγνωρίσει. Όλα αυτά μας κάνουν να σκεφτούμε πώς θα ασκήσουμε πιέσεις στο Βελιγράδι. Καμιά φορά αυτό οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα και απομακρύνουμε ένα μέρος του πληθυσμού του κοσμοπεδίου από την Ευρώπη. Σχετικά με την παράγραφο 9, με την, σχετικά με την EULEX, καλούνται τα κράτη ε, που ανήγγυλαν ε, την απόσυρση των αστυνομικών δυνάμεων ε, καλούνται να σκεφτούν το θέμα αυτό. Σχετικά με την κατάσταση της Ρουμανίας που το ανήγγειλε αυτό, νομίζω ότι υπάρχει συνένεση για το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, και αυτό είναι ενημερωτικό, να επανεξετάσει την απόφασή της η Ρουμανία. Δεν υπάρχει καμία υποστήριξη για μια τέτοια μεταστροφή. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να παραδεχθώ ότι είμαι κάπως απογοητευμένη με το κείμενο της κυρίας Λούνατσέκα διότι η συγγήτρια φαίνεται να μην δέχεται την πραγματικότητα ότι πέντε κράτη-μέλη δεν έχουν αναγνωρίσει τη χώρα αυτή. Και πάντως αυτή η εισήγηση δεν μπορεί να είναι ένα μέσο άσκησης ε, εξουσίας ή πίεσης για να αναγνωρίσουν οι χώρες αυτές το κοσμοπέδιο. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Εμείς τι θέλουμε εμείς ο Κοινοβούλιο. Θέλουμε να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα στον πληθυσμό του Κοσμοπεδίου ότι έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική. Γι' αυτό η πλειονότητα ημών υποστηρίζει την απελευθέρωση, σχετικά και, ότι, χαιρόμεθα που θα αρχίσει ο διάλογος για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Ελπίζω ότι αν επιτύχουμε αυτό το στόχο θα είναι ένα θετικό μήνυμα, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα κράτη-μέλη που έχουν νομικές και πολιτικές αντιρρήσεις δεν θα αλλάξουν τη θέση τους εκτός αν βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για το θέμα του καθεστώτος του Κωσυφοπεδίου. Το δεύτερο σημείο μου είναι ο διάλογος ανάμεσα στην Πρίστινα και στο Βελιγράδι. Θα πρέπει να επανεξισορροπήσουμε το κείμενο, διότι διαβάζοντας το κείμενο ως έχει, πέφτει όλη η ευθύνη πάνω στο Βελιγράδι. Όπως περιγράφεται ως άμεσο αποτέλεσμα, ε, μη υλοποίηση συμφωνιών κλπ. Και παραβλέπετε το γεγονός ότι ήταν η αστυνομία του Κοσφοπεδίου που πυροδότησε την κρίση πέρσι. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε μια νέα παράγραφο 6 σχετικά με την απόφαση του Βελιγραδίου να ξαναρχίσει τον διάλογο με την Πρίστινα. Αλλά πάντως η θέση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι να καδεκατικάσει οποιοδήποτε διάβημα, οποιοδήποτε διάβημα μονομερές, οποιοδήποτε αποκλεισμό ή χρήση βίας είτε προέρχεται από τη σερβική πλευρά είτε από την πλευρά των Κωσοβάρων. Τέλος, η ευρωπαϊκή προοπτική είναι σημαντικό στοιχείο μέσα σε αυτό το πλαίσιο και θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι ο μόνος διάλογος Μόνο διάλογος είναι ο τρόπος ε, για να προοδεύσουν και να ευημερήσουν όλοι οι πολίτες ε, της περιοχής, όλοι οι κάτοικοι. Η απόφαση να δοθεί καθεστώς υποψηφίας χώρα στο Κωσυφοπαίδιο είναι κάτι το οποίο διακυβεύεται. Η πίεση είναι από την πλευρά του Βελιγραδίου. Θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο την ανάγκη οι αρχές της Πρίστινα να σέβονται τα θεμελιώδη ε, δικαιο... ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους πολίτες και να ζητήσουμε από τις αρχές να προσπαθήσουν ούτω ώστε οι Σέρβοι του Κοσφοπεδίου να αισθάνονται ασφαλείς και να μην υποχρεώνονται να φύγουν από τις αιστείες τους. Ευχαριστώ την κυρία Κοπά. Ο κύριος Μπρόκ για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Νομίζω ότι έχει γίνει αρκετά σαφές ότι το κοσφοπέδιο δεν έχει αναγνωριστεί από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ακόμα επίσης εσωτερικά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν για να γίνει λειτουργικό κράτος το κοσφοπέδιο. Υπάρχει το θέμα της εσωτερικής ε, ανάπτυξης, του νομικού συστήματος. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διοίκηση, αλλά φυσικά και με την διαφωνία, τη διαμάχη με την ε, Σερβία. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε πρόοδο, αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι εάν κάποια στιγμή το κοσμοπέδιο εκπληρώσει τα απαιτούμενα, θα μπορέσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κεφαλαιόδες για να εξασφαλίσουμε την σταθερότητα της χώρας αυτής. Οι συζητήσεις στην ε, Θεσσαλονίκη για τη σταθερότητα της περιοχής είχαν σαν στόχο να επιτύχουν ακριβώς αυτό το στόχο. Και η εμπειρία μας από τα χρόνια του πολέμου είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να υπερκεραστούν οι διαμάχες και οι συγκρούσεις του παρελθόντος χωρίς μια τέτοια προοπτική. Επομένως, αυτό είναι ένα βασικό θέμα, αν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις κατά πόσο θα είναι θετική ή όχι η, η είσοδος του κοσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέτε ότι κοστίζει πολύ. Μα όλοι οι μηχανισμοί σταθερότητας, όλοι οι μηχανισμοί ασφάλειας κοστίζουν λεφτά και οι στρατιώτες κοστίζουν λεφτά. Όταν χύνεται αίμα στην Ευρώπη, αυτό κοστίζει ακόμα περισσότερο. Μπορεί ο Dartmouth να αναφέρεται σε αυτοκρατορικά σενάρια και οράματα, αλλά στην πραγματικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε σε αυτή την περιοχή που πάντα ήταν περιοχή αστάθειας και έχει αποτελέσει και την απαρχή και το έναυσμα πάρα πολλών πολέμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσουμε μια γαλήνη. Λοιπόν, το να ονομάζει κανείς κάτι τέτοιο μια μορφή αυτοκρατορικών σενάριων και οραματών, αυτό δείχνει ότι δεν έχει την πνευματική ικανότητα να κατανοήσει πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω σε σχέση με την εκθέση της κυρίας Λούνατσεκ ότι όταν αναφέρεται το κοσυχοπαίδιο δεν αναφέρει η συγγήτρια και το ψήφισμα των, του Συμβουλίου Ασφαλείας ούτε καν και τα έγγραφα τα οποία περιλαμβάνουν μια μνήα στο, στην απόφαση αυτή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στην παράγραφο 1 λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χαιρέτιζε το να δεχτούν τα πέντε ακόμα κράτη που δεν το έχουν δεχτεί να δεχτούν τη μονομερή ανεξαρτησία του Παιδί, Αυτό σημαίνει ότι επιμένει η συγκίτρια σε μια θέση για ένα θέμα το οποίο δεν είναι στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σίγουρα οδηγεί σε διχασμό μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί ο στόχος μας εδώ θα έπρεπε αντίθετα να είναι να έχουμε μια ως τον ετών πιο ενωμένη θέση. Στην παράγραφο 6 θεωρεί υπεύθυνη τη Σερβία γιατί δεν έχει εφαρμόσει τις ε, συμφωνίες οι οποίες είχαν συναυθεί και ζητάει από τη Σερβία να κάνει τα απαραίτητα βήματα για να μπορέσει να υπάρξει επαναφορά του διαλόγου. Εδώ πρέπει να το διαφοροποιήσουμε αυτό. Γιατί η Σερβία ήταν αυτή η οποία έφερε το ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη. Η Κομισιόν έχει αναγνωρίσει στην τελευταία της ανακοίνωση το ότι η Σερβία έχει πράγματι λάβει τα πρώτα μέτρα για να εφαρμόσει το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών και η Εντίτα Τάιρη η διαπραγματευτή του Κωσόβου δέχεται ότι η Σερβία έχει εφαρμόσει τη Συμφωνία Ελευθερών Εμπορίου. Λοιπόν, είναι υπερβολικό να πούμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί καμία συμφωνία. Η θέση των χωρών που δεν έχουν δεχθεί το κοσυφοπέδιο, το έχουν αναγνωρίσει το Κωσυφοπέδιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι είναι μια σόφρον θέση που ενισχύει τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό επέτρεψε να υπάρξουν συζητήσει υψηλού επίπεδου Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκανίων που υποστηρίχθηκαν στο εξάμεινο της Ισπανικής Προεδρίας, όλα αυτά οδήγησαν σε μια ομόφωνη έγκριση του ψηφίσματος Σεπτεμβρίου 2010 από την ε, Σερβία και την, ε, τα Έθνη σε σχέση με ένα διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας και συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Αν όλα τα κράτη-μέλη λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν μονάχα τη μία πλευρά, υποστηρίζουν τη μία πλευρά, αυτό ο διάλογο μάλλον δεν θα ήταν εφικτό. Και θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να απορρίψει την προσπάθεια να επιτύχει μια ευρεία συνένεση σε σχέση με το καθεστώς του Κωσυφοπεδίου. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε και την διεθνή νομιμότητα διατηρώντας τον επίσημο τίτλο του Κωσυφοπεδίου και να αφήσει στα κράτη-μέλη να, μέσα στην κυριαρχία τους το μέλημα του να αναγνωρίσουν ή όχι ένα κράτος όπως το Κοσμοπέδιο, γιατί αυτό είναι υπόθεση των κυριαρχών κρατών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στο κοσφοπέδιο και επηρεάζουν τους πολίτες αυτής της χώρας και να επιληθούν πολλά από τα προβλήματα τα οποία αναφέρονται και στην ανακοίνωση της Κομισιόν και στο σχέδιο της ε, εισηγήτριας, οργανωμένο έγκλημα, κράτος δικαίου, δικαστική εξουσία, δημόσιος τομέας, οικονομική κατάσταση και όχι σε ζητήματα να εστιάσει η έκθεση αυτή που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω διαμάχηση μέσα στο Κοινοβούλιο. η επανάληψη των συζητήσεων στην Πρίστινα νομίζω ότι θα βοηθήσει την προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών. Και θέλω επίσης να τονίσω ότι και από την πλευρά του Συμβουλίου υπήρξε μια ανακοίνωση όπου αναγνωρίζεται η επανάληψη του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών. Ε, Κοιτάξτε, εγώ δίνω το λόγο σύμφωνα με ένα αυστηρό κριτήριο. Πρώτα δίνω το λόγο στους και όλους εφόσον είναι παρόντες. Μετά παίρνω τη χρονολογική σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τα πολιτικά κόμματα έκανα ένα λάθος με τον κύριο Αυλάκη γιατί θυμόμουν ότι ήταν στην ελεύθερη ομάδα ενώ έχει περάσει σοσιαλιστές. Βάση περιπτώσει αυτό ε, δεν το έκανα σαν λάθος. Αυτοί είναι οι κανόνες μου λοιπόν. Εγώ δεν έχω προτιμήσεις για ονδήποτε. Εσείς μπορείτε να ερμηνεύσετε βέβαια αυτό που κάνω με διαφορετικό τρόπο. Κύριε Βότσον. Εσείς φτάσατε τελευταίος, παρόλα αυτά δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ένα λεπτό παρακαλώ, άντε δύο λεπτά το πολύ κύριε Βότσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα παραμείνω μέσα σε ένα λεπτό, έτσι κι αλλιώς δεν περίμενα να πάρω το λόγο, αλλά δεν υπάρχει κανείς από την ομάδα μου θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζουμε πλήρως την ισόρροπη γενικά αντίληψη που εκφράζει η έκθεση αυτή. Η συγγήτρια έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Νομίζουμε ότι το κοσυφοπαίδιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί δίκαια όπως όλες οι άλλες χώρες. Είναι μια νέα χώρα, αλλά παρότι νεαρή χώρα ξεπέρασε τη συνταγματική κρίση που αντιμετώπιζε επιτυχώς και νομίζω ότι οι προτάσεις της εισηγητρίας είναι σωστές και θα τις στηρίξουμε. Ευχαριστώ κύριο Βότσον και για την συνθετικότητά σας. Τα τελικά σχόλια, όχι πάνω από τρία λεπτά, παρακαλώ η κυρία Λούνατσεκ. Θα προσπαθήσω μέσα σε τρία λεπτά. Εν πάση περιπτώσει θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ευχαριστώ και αυτούς οι οποίοι υποστήριξαν την έκθεση, όπως οι τελευταίοι ομιλητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και αυτούς που άσκησαν κριτική σε αυτά τα οποία λέγω και το ήξερα αυτό. Να αναφερθώ μου σε κάποια από τα θέματα τα οποία έφτιαξαν οι τελευταίοι. Αυτό το οποίο πολλοί από σας επαναλάβατε είναι η κριτική η οποία γίνεται σε σχέση με το Ulex. Ε, ξέρω ότι έχει ασκηθεί κριτική και στο παρελθόν στη Ulex θα ήθελα να προσπαθήσω να δω τι είδους πληροφορίες μπορούμε να συλλέξουμε γύρω από την λειτουργία της γιουλέξ. Παρ' όλα αυτά είμαι βέβαιος ότι στα πλαίσια της εντολής την οποία θα πρέπει να έχει η γιουλέξ απαιτείται να υπάρξουν ορισμένε μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι ήδη στο pipeline. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με αυτούς οι οποίοι στηρίζουν τη Ulex. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας εδώ και με τους άλλους και όλους συγητές. Να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ντάθμαουθ για τη σημασία των μέσων ενημέρωσης. Λοιπόν, τι σας λέω, μία λέξη, Μέρντοχ. Λοιπόν, α, δεν με ακούει γιατί δεν είναι εδώ ο κύριος Ντάθμαουθ. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν σκάνδαλα πάρα πολύ, ε, περισσότερα σκάνδαλα διέπραξε ο συγκεκριμένος κύριος ε, από ότι η ίδια η χώρα του Κωσυφοπεδίου. Λοιπόν, τώρα, να αναφερθώ σε συναδέλφους οι οποίοι άσκησαν ε, κριτική και προέρχονται από χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει τη χώρα. Κοιτάξτε, μια αντίστοιχη διατύπωση έγινε δεκτή και πέρυσι με μεγάλη πλειοψηφία. Γνωρίζω τις θέσεις των χωρών αυτών και των κυβερνήσεων αυτών των χωρών. Κάποιες κυβερνήσεις αλλάζουν σε αυτές τις χώρες. Ίσως να υπάρξει μια αλλαγή στη θέση τους. Λοιπόν, νομίζω ότι εμείς ε, δεν εκφράζουμε εδώ τις θέσεις των χωρών μας, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση του κοσφοπεδίου είναι ευρωπαϊκό θέμα. Και υπάρχουν βέβαια ε, κάποιες, ε, κάποιες από αυτές τις χώρες εσωτερικά θέματα που εμποδίζουν την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του κοσφοπεδίου. Ελπίζω όμως να πετύχουμε για μια ακόμη φορά μεγάλη πλειοψηφία για κάποια κριτική που ασκήθηκε για την πρόοδο στο Κοσφοπέδιο. Κοιτάξτε και κάνω κάποια κριτική για το ότι δεν έχει πετύχει το Κοσφοπέδιο. Απαιτείται περισσότερη πρόοδο στο Κοσφοπέδιο. Of my uh, here and if you read it well... Λοιπόν, αν διαβάσετε προσεκτικά την έκθεσή μου θα ικανοποιηθείτε. Για τον κύριο Τάνοκ, εξεπλάγει όταν είπατε ότι το Κοσφοπέδιο γίνεται μια μονοπολιτιστική χώρα. Δεν ξέρω σε ποια χώρα έχετε πάει στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα δείτε μέλη του Κωσυφοπεδίου να προέρχονται από την αλβανική πλειοψηφία αλλά και από τους Σέρβους και από τους Ρωμά και από τους Αιγυπτιογενείς και γενικά από όλους αυτούς οι οποίοι συνθέτουν ε, το κοινοβούλιο. Πού τη βλέπετε τη μονοπολιτιστική πλευρά του Κωσυφοπεδίου για τη σερβική μειονότητα Ξέρετε κύριε Τάνοκ ότι και στον Νότο υπάρχουν δήμαρχοι, υπάρχουν δήμοι, σερβικοί, στο Βορρά υπάρχει θέμα και αναφέρομαι σε αυτό. Ελπίζω ότι ο διάλογος θα οδηγήσει σε κάποια θετική κατάληξη. Βλέπω βέβαια ότι η Σερβία θα χρειαστεί να εφαρμόσει κάποιες νέες αποφάσεις. Ε, άκουσα τις δηλώσεις της κυβέρνησης, ξέρω ότι υπήρξαν ήδη κάποια σημεία προόδου σε σχέση με τους τίτλους, αλλά παρόλα αυτά απαιτούνται περισσότερο, περισσότερα βήματα και εγώ είμαι υπέρ της απόδοσης του τίτλου της υποψηφίας χώρας στη Σερβία, αλλά το ίδιο πρέπει να γίνει και το κοσφοπέδιο, όπως έχει πει και ο Επίτροπος Φούλε. Η προσθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 13η Δεκεμβρίου, θα τα Λοιπόν, η συζήτηση των τροπολογιών θα γίνει στις 23-24 Ιανουαρίου και η ψηφοφορία επίσης. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε σε μια πρόταση σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για τους τρόπους της πιθανής δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Δημοκρατία. Είναι η πρώτη συζήτηση η οποία γίνεται εδώ. Θα σας παρακαλέσω να είσαστε πάρα πολύ σύντομοι. Ε, θα έχουμε σε μια άλλη φάση την συζήτηση σε βάθος και περιμένουμε σε 7 λεπτά τον Σέρβο Υπουργό. Γι' αυτό παρακαλώ ε, μπορέστε να είστε σύντομοι για το ευρωπαϊκό κληροδότημα για τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε συζητούμε πράγματι αυτή την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο για, τους, για τις ε, λεπτομέρειες και τις διατάξεις σε σχέση με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ε, κληροδοτήματος για τη δημοκρατία. Έχουν δείξει οι εξελίξεις στην, στον αυρικό κόσμο και αλλού ότι τα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη της δημοκρατίας δεν είναι επαρκή για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες και θα ήταν χρήσιμο να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ε, πραγματικές καταστάσεις και να μπορεί να έχει ταχεία αντίδραση όταν χρειάζεται. Είναι φανερό ότι η Προεδρία, η τωρινή Προεδρία υποστηρίζει ιδιαίτερα το σχέδιο αυτό και έχει έρθει σε επαφή με τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν δεχτεί την καταρχήν δημιουργία ενός τέτοιου ταμείου στις 20 Ιουνίου του ενεστώτος έτους. Στη δική μας σύσταση η οποία προέκυψε μετά από πολλές συζητήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές και με μια επίσημη συνάντηση όλων των εισηγητών και συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Υπήρξε συζήτηση η οποία περιλαμβάνει τις θέσεις όλων των πολιτικών ομάδων. Έχουμε καταλήξει σε ορισμένε θέσεις, οποίες θα παρουσιάσω εν συντομία και ελπίζω ότι αν υπάρχουν ερωτήσεις μπορούμε να επανέλθουμε. Καταρχήν, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνει το ταχύτερο δυνατό αυτό το, αυτό το ταμείο για να υποστηρίξει τη βαθιά και βιώσιμη δημοκρατία. Πρόκειται για χώρες οι οποίες βρίσκονται σε μια διαδικασία καμπής ή αλλαγής, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες εταιρικέ σχέσεις με φορείς και δυνάμεις στις χώρες αυτές. Είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να επιδιώξουμε να έχουμε και τέτοιου είδους εταιρικές σχέσεις με άλλες χώρες οι οποίες υποστηρίζουν τη δημοκρατία και με τα δικά τους Ινστιτούτα ή τους δικούς φορείς, αλλά φυσικά και με το Ευρωπαϊκό Μέσο για Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα συμπληρωματικό ρόλο και να εξασφαλίσουμε συνέργειες. Να έχουμε λοιπόν ένα ταμείο το οποίο θα δίνει χορηγήσεις, θα μπορεί χρηματικά να δίνει υποστήριξη, αλλά το οποίο δεν θα είναι παρόν σε λειτουργικό επίπεδο επί το θα μπορεί να ενισχύσει σχέδια σε διάφορες χώρες με τη βοήθεια εταίρων οι οποίοι θα βοηθήσουν στην εφαρμογή ακολουθώντας το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ αυτού του Ταμείου και του Ταμείου για την Δημοκρατία. Οι φορείς λοιπόν εδώ πέρα, οι πέκτες που θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιγραφούν με έναν τρόπο ο θα είναι σαφής. Το ουσιαστικό είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε εταίρους και παίκτες οι οποίοι για νομικούς ή άλλους λόγους δεν μπορέσανε μέχρι στιγμής να υποστηριχθούν από το μέσο για τη δημοκρατία. Δεν πρόκειται για κομματική υποστήριξη, δεν πρόκειται για προώθηση μιας πολιτικής ατζέντα με, κομματική, με κομματικές πτυχές. Αντίθετα, είναι να δώσουμε σε ορισμένε πολιτικές δυνάμεις τη δυνατότητα να παίξουν κάποιο ρόλο στα τεκτενόμενα της ε, χώρας τους. Θα έχουμε λοιπόν μια δομή η οποία θα βρίσκεται στην Βρυξέλλες θα μπορεί να παίρνει πληροφορίες από τα γεωγραφικά γραφεία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και θα έχει και μία δομή διακυβέρνησης, όπως προέκυψε από την ε, διαβούλευση, ώστε να εξασφαλίσει ότι τα ευρωπαϊκά αυτά κονδύλια θα είναι ελέγξιμα και υπόλογα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξασφαλιστεί και μια πολιτική υποστήριξη. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει μια θέση η οποία δεν θα εξασφαλίζει αυτή η πολιτική ισορροπία και σας ευχαριστώ και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Λάντστορφ. Η κυρία Σαϊφή, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Λάμπστορφ ε, για την, ε, τις παρατηρήσεις του και είχαμε την δυνατότητα να ανταλλάξουμε ιδέες για το θέμα αυτό. Βεβαίως τα όσα συνέβησαν στον αραβικό κόσμο πρόσφατα μας οδηγούν στο να αναθεωρήσουμε την στρατηγική συνεργασία με όλες αυτές τις χώρες. Η δημιουργία αυτού του κληροδοτήματος θα πρέπει να αποφέρει μια πραγματική προστιθέμενη αξία στα προγράμματα βοήθειας προς τις μελλοντικές δημοκρατίες. Θα πρέπει να είναι μια ελαφρά ε, δομή και μια όχημα ε, απλουστευμένης χρηματοδότησης ε, επιτρέποντας μια μεγαλύτερη αντιδραστικότητα και ευελιξία. Θα πρέπει να επιτρέπει μια μεγαλύτερη προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της δημοκρατίας ενώ θα πρέπει να αποφύγουμε να μην κατηγορηθεί η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση για ανάμειξη στα εσωτερικές υποθέσεις των γειτόνων. Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Η πρώτη, διερωτώ με για τη σκοπιμότητα ενός ε, μιας χρηματικής στήριξης από το κληροδότημα στα πολιτικά κόμματα. Ποιες θα είναι οι εγγυήσει που θα έχουμε. Δεν υπάρχει κίνδυνος η ουδετερότητά μας και η ισορροπία που θα πρέπει πολλές φορές να διαφυλάξουμε να θίγονται. Δεν θα ήταν πιο σκόπιμο να δείσουμε ιδρύματα ή μη κυβερνητικέ οργανώσεις ούτως ώστε οι δράσει Ευρωπαϊκής σαν να μην θεωρείται προσπάθεια ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις μιας χώρας. Δεύτερη παρατήρηση. Το κληροδότημα αυτό θα πρέπει σε μια πρώτη φάση να υποστηρίζει την μετάβαση, την δημοκρατική των ε, γειτόνων μας. Η ζώνη γεωγραφική του κληροδοτήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του κόσμου, αλλά να αποδίδει ιδιαίτερη ε, σημασία κυρίως για στα μελλοντικά χρόνια στους γείτονες οι οποίοι είναι πιο κοντά στην Ευρώπη. Άλλη παρατήρηση, το κληροδότημα αυτό θα έπρεπε όπως γίνεται ε, σε μερικά κράτη-μέλη τώρα να χρηματοδοτεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ε, πρόσκλησης ε, μελλοντικών προσωπικότητων που εμπλέκονται άμεσα στην προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό θα επέτρεπε να διευκολύνουμε την επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτάσσοντας γυναίκες και άνδρες που εργάζονται για την δημοκρατία. Τελευταία παρατήρηση σε σχέση με την διοικητική μέθοδο για να ελαφρύνουμε όσο το γίνεται περισσότερο την διακυβέρνηση ε, και τα έξοδα διαχείρισης. Ποια είναι η δομή που θα ήταν η πιο σκόπιμη, ένα ίδρυμα ή ένα εικονικό ταμείο. Ε, θα μπορούσε αυτό να συνδέεται διοικητικά με την ε, Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ούτως ώστε να υπάρχει συνεκτικότητα με την συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως και κλείνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνδεθεί στενά με την υλοποίηση, την διαχείριση και έλεγχο αυτού του κληροδοτή μας. Κυρία Γκόμες, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάω εξ ονόματος της Βερονίκλουπες που είναι σκιώδης η για την ομάδα μας. Δεν μπόρεσε να είναι εδώ και μου ζήτησε να λάβω τον λόγο στο όνομά της. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα διότι ήμουν από τους πρώτους που χαιρέτησαν την ιδέα της δημιουργίας ενός τέτοιου ε, κληροδοτήματος ε, το 2010 και αυτό διότι αισθάνομαι την ανάγκη να υπάρχει ένα τέτοιο κληροδότημα. Η Βερονίκα μου ζήτησε ένα. Ε, ότι να υποβάλω το θέμα ότι ο έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η υποπτία είναι κάτι το σημαντικό στις στρατηγικές της χώρας, στον έλεγχο της διαχείρισης. Θα έπρεπε το Διοικητικό Συμβούλιο, την σύνθεση να εξεταστεί, να μην είναι αυτή των κατευθυντηρίων γραμμών, δεν θα είναι μια δομή γραμμική όπως αναφέρουν οι κατευθυντήριες γραμμές που εξετάζει το Συμβούλιο βάσει των ιδεών που αναπτύχθηκαν, όπως προβλέπετε σε αυτές, διότι θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε κράτο ε, μέλος που ε, συμβάλλει, θα μπορούσε να είναι μέλος. Αλλά δεν θέλουμε τέτοια βαριά δόμη. Θέλουμε καλύτερη εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου που να αντικατοπτρίζει όλο το πολιτικό φάσμα αυτού του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα για να μπορεί να λειτουργεί καλά αυτό το Ταμείο για αυτά τα οποία πρέπει να κάνει, δηλαδή τη στήριξη της ε, δημοκρατίας παντού στον κόσμο. Ένα άλλο στοιχείο είναι μια εκπροσώπηση πολιτικά εξισορροπημένη με εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου βεβαίως που να εκπροσωπεί όλο αυτό το φάσμα. Και η Βερονίκ πιστεύει ότι η κατανομή ε, πόρων και κονδυλίων ε, θα πρέπει να γίνει σε πρωταγωνιστές επιτόπου και όχι μεταξύ Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων. Αυτό και θα, ε, πρότεινε και ο Αλεξάνδρ και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την δουλειά του. Θα προσθέσω τα δικά μου σχόλια. νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παράγοντες, αυτούς που είναι δραστήριοι επιτόπου ή μπορούν να γίνουν δραστήριοι επιτόπου θα, μπορεί να είναι πολιτικά κόμματα, μπορεί να είναι ιδρύματα. Δεν πρέπει λοιπόν να τους παραβλέψουμε. Δεύτερη ερώτηση, τελευταία ερώτηση. Ε, πώς προβλέπεται η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι από το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αντληθούν τα κονδύλια. Όχι, όχι, εκεί δεν υπάρχει πολλή χρηματοδότηση και έχει αντίκτυπο πάνω στην προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βεβαίως, αλλά πρέπει να πάρουμε χρήματα από αυτούς που δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως θα έπρεπε να είναι DCI, ICI. Ε, αυτό εξαρτάται από την ε, γεωγραφική περιοχή ε, όπου βρίσκονται και δεν πρέπει να περιορίζονται στην γειτονία, στις γείτονες. Ευχαριστώ. Λοκ Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαβάσαμε το σχέδιο έκθεσης, το θεωρώ θετικό, αλλά είναι κάπως δύσκολο να έχουμε σαφείς όρους αναφοράς για αυτό το κληροδότημα. Γιατί βλέπουμε ότι ακόμα δεν είναι σαφείς οι όροι αναφοράς. Εμείς θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε αυτό να είναι σαφές ήδη από την απαρχή αυτής της διαδικασίας, τουλάχιστον να έχουμε μια αδρή ιδέα για τη μορφή αυτού του κληροδοτήματος. Θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, ε κόμιτα Λάμστορφ αν αυτό θα έχει κάποια αποτελέσματα, κάποια επιρροή στο ψήφισμα, το γεγονός ότι ακόμα δεν είναι σαφή τα βασικά, οι γενικές γραμμές αυτού του κληροδοτήματος. Νομίζω ότι παραμένουν ακόμα πολλά ανοιχτά ερωτήματα ως εκ τούτου. Για μας ως πράσινους είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε καταθέσει σχετικά τροπολογίες να υπάρξει συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Είπαμε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν μάλλον χρησιμοποιηθεί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει αυτό το ίδρυμα, θα πρέπει να γίνει με τρόπο που συνάδει με το δημοσιονομικό κανονισμό και γι' αυτό θα θελήσουμε και πάλι με μια τροπολογία να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει περαιτέρω πάνω από 50% χρηματοδότηση αυτού του κρυοδοτήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπορούμε να τροποποιήσουμε τη διατύπωσή μας ότι δεν θα πρέπει, ζητούμε σε μια τροπολογία, να μην υπάρξουν περαιτέρω περικοπές στο μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλληλοεπικάλυψη των δύο αυτών ταμείων. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το κλειοδότημα για θα πρέπει να αντιμετωπίσει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου υπάρχουν ήδη σχέδια της υπάρξης αρμοστίας για τους πρόσφυγες και τα λοιπά και του μέσου για τη δημοκρατία. Θέλουμε να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτό το μέσο με τις προϋποθέσεις που ανέφερα. Ευχαριστώ κυρία Λόχμπιχλερ. Κλείνει τη συζήτηση κύριος Λέσσινγκ δύο λεπτά. Η κυρία Λέσσινγκ, συγγνώμη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ομάδας μου μπορώ να πω ότι εμείς αντιμετωπίζουμε με μεγάλο σκεπτικισμό αυτό το εργαλείο και βλέπουμε σημαντικά ελλείμματα δημοκρατία. Αυτή συγκεκριμένα η φιλοδοξία να υπάρχει ταχεία αντίδραση από αυτό το μέσο, για μας είναι κάτι το οποίο δεν μας ικανοποιεί και θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και ενίσχυση στο μέσο αυτό. Θεωρούμε ότι αυτό το ε, μέσο καταρχήν δεν μας ικανοποιεί, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία να κάνουμε ορισμένε προτάσεις για να βελτιώσουμε την επεξεργασία του. Έχει ήδη αναφερθεί το ένα από αυτά τα θέματα. Θα ήθελα Ναι, ναι, δεν θα σας τα διαβάσω, θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη. Δίνουμε μεγάλη σημασία στο να τηρηθεί η αρχή της κυριαρχίας και να μπορέσει αυτό το εργαλείο να μην χρησιμοποιηθεί, να μην τύχει καταχρήσεως για να εξυπηρετήσει άλλα συμφέροντα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει ο έλεγχος του προπολογισμού και ο κοινοβουλευτικό έλεγχος και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο πριν δοθούν τα χρήματα αυτά να υπάρξει κάποιος ανώτερος φορέας ο οποίος θα είναι σε θέση να ελέγξει τη χρηματοδότηση αυτή και να υπάρξει κάποιο έλεγχο για το σε ποιου δίνονται και πώ δίνονται αυτά τα χρήματα. Eh, Ευχαριστώ κύριε Λόζινγκ. Ζητώ συναδέλφοι από του συναδέλφου Πρέντα και Σαβλουσβόλσκι και κάποιον άλλον που δεν άκουσα το όνομα. Δεν μπορώ να του δώσω το λόγο. 8 Δεκεμβρίου όταν γίνει η κανονική συζήτηση μα περιμένει ο κύριο Υπουργό αν ο κύριος Λάμπσδορφ θέλει να κάνει τρία, εισαγω, λεπτά εισαγωγικά σχόλια, αλλά όχι περισσότερο παρακαλώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι για αυτά που μου ανέφεραν οι συνάδελφοι. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά στοιχεία. Υπάρχει καταρχήν μια ευρεία συνένεση μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω της μορφής αυτού του Ταμείου δεν θα πρέπει όχι μονάχα να έχει και, και έλεγχο ως θεσμικός φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως δημοκρατικά εκλεγμένος φορέας να εξασφαλίσει ότι θα κατευθύνεται προς τη συγκεκριμένη αυτή κατεύθυνση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα καταγραφεί φυσικά στην έκθεση. Υπάρχουν ορισμένα σημεία ακόμα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε και θα πρέπει να συζητήσουμε για όλα αυτά. Όταν λέει η Βερονίκ Δικεζέρ ότι θα πρέπει τα χρήματα αυτά να πάνε σε τοπικούς παίκτες. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό με μια ευ ελαφρύ δομή στις Βρυξέλλες χωρίς την επιτόπια γνώση που θα μας δώσουν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις όπως η ΜΚΟ επιτοπίως. Αυτό επίσης το ερώτημα το οποίο έθεσε η Μπάρβαρα Λόχλερ ότι δεν πρέπει να υπάρχει παραπάνω από 50% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην επηρεάσει ιδιαίτερα την εσωτερική στάθμιση. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι λοιπόν να επιλύσουμε όλα αυτά τα θέματα και επίσης η κυρία Σαΐφη τόνισε το εξής ερώτημα με ποια μορφή θα επιλέγουμε αυτούς τους πολιτικούς εταίρους. Είπαμε σαφώς ότι δεν θέλουμε να έχουμε χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, αλλά πολλές φορές κινήματα, πολιτικά κινήματα που βρίσκονται στον περίγυρο ε, πολιτικών κομμάτων, όταν παραδείγματος χάρη υπάρχει Υπάρχουν για πρώτη φορά ελεύθερε εκλογέ ή κινήματα τα οποία προσπαθούν να σφυριλατήσουν ορισμένε κατευθύνσει. Εκεί θα πρέπει να κάνουμε μια στρατηγική εκτίμηση που θα πρέπει να είναι αντικείμενο κοινή συζήτηση και να δούμε ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να επιλύσουμε τέτοια θέματα. Και το τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω, η Μπάρμπαρα Λοχμπίτερ έθεσε επίση το θέμα του ότι δεν είναι ακόμα σαφή η όρια αναφορά. Προβλέπετε την 1η Δεκεμβρίου προβλεπόταν 1η Δεκεμβρίου να υπάρξει ο καθορισμός των όρων αναφοράς, τώρα ουσιαστικά έχει αναβληθεί αυτή, αυτός ο καθορισμός, αλλά έχω προτείνει ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα, ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να συζητήσει για τα θέματα αυτά. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα αν υπάρξει αλλαγή των όρων αναφοράς. Θα πρέπει να τροποποιηθεί η προθεσμία για τις τροπολογίες, ώστε να μπορέσουμε να ε, κάνουμε τις δικές μας ε, αλλαγές στις συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταίο σημείο, υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον από αυτά που είπε η κυρία Σάιφη, να υποστηρίξουμε προσωπικότητες του μέλλον, δηλαδή να υποστηρίξουμε ανθρώπους που είναι νέοι και έχουν δυναμικό για το μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να το κάνει αυτό. Λόγω της ώρας ε, θα κλείσω εδώ και μπορούμε να συζητήσουμε και άλλη μια φορά. Αύριο έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας να ζητήσει για το θέμα αυτό και αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ κύριε Λάνσδορφ. Όπως ξέρετε επαναλαμβάνω στις 8 Δεκεμβρίου θα γίνει η πρώτη θα έλεγα σε βάθος συζήτηση της προτάσεως. Η σημερινή συζήτηση ήταν απλά προκαταρτική περιμένοντας τον Πολωνό Υπουργό αύριο. Προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών θα είναι η 15η Δεκεμβρίου και για τη συζήτηση και την ψηφοφορία το επόμενο Φεβρουάριο. Το επόμενο θέμα είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Βούκ Τζέρεμιτς, Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας, ο οποίος μπορεί να εισέλθει τώρα. Buongiorno. Possiamo... Καλημέρα σας. Καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Τζέρεμιτς. Ο κύριος Γέρεμιτς είναι υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας. Τον καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά. Εκφράζουμε εξ ονόματος όλων τα συγχαρητήριά μας για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στο Συμβούλιο να δώσει στην χώρα σας το καθεστώς της υποψηφίας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια σαφέστατη αναγνώριση και ένα κίνητρο για τις διαδικασίες της μεταρρυθμιστικές τις οποίες έχει ήδη εν μέρη ολοκληρώσει η χώρα σας αν και σίγουρα υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα για να μπορέσουμε να διανύσουμε τον σύνολο δρόμο που θα οδηγήσει στην κατάληξη της πορείας που από κοινού ξεκινήσαμε. Πάντως ελπίζουμε ότι τον μήνα Δεκέμβριο το Συμβούλιο θα υιοθετήσει τη σύσταση της Κομισιόν. Το καθεστώς της υποψήφιας χώρας, όπως γνωρίζετε, συνδέεται με μία προϋπόθεση, την βελτίωση στη συγκεκριμένη περίπτωση των σχέσεών σας με το κοσφοπέδιο. Το είδαμε και στη συζήτηση η οποία προηγήθηκε. Ε, πρόκειται για ένα πρόβλημα καμφόδες, για ένα πρόβλημα ευαίσθητο, ένα θέμα το οποίο απαιτεί όμως και μια πραγματιστική και συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι ο διάλογος με την Πρίστινα που ξεκίνησε τον προηγούμενο Μάιο συνεχίζεται. Υπήρξαν αρκετά σημαντικές θα έλεγα συμφωνίες σε ορισμένα συγκεκριμένα σενάρια, αλλά παρόλα αυτά οι συνθήκες συμβίωσης των κοινοτήτων της Σερβίας, των Σερβικών και των Αλβανικών δεν έχουν θα έλεγα φτάσει στο κατάλληλο επίπεδο. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει και σε άλλα υπάρχει μια σαφέστατη επιβράδυνση. Υπήρξε μια πρόσφατη συνάντηση από την οποία προήλθε μια συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων, αλλά παρόλα αυτά θα έλεγα δεν έχει καταλήξει η διαδικασία ακόμη εκφράζω την ευχή κάτι τέτοιο να γίνει. Ελπίζω να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα και άλλα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Δεν θέλω να σας κλέψω περισσότερο χρόνο. Σας δίνω αμέσως το λόγο και θα σας ακούσω με πάρα πολύ ευχαρίστηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέτετε και σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ να συζητήσετε το ευρωπαϊκό μέλλον και την ευρωπαϊκή προοπτική για το σύνολο των Δυτικών Βαλκανίων αρχίζοντας από τη Σερβία. Ξέρω ότι είναι δύσκολη εποχή στην Ευρώπη και υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα που συζητούνται ίσως πιο άμεσου ενδιαφέροντος για τους λαούς που σας έχουν εκλέξει. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων για το χρόνο που μου αφιερώνετε σήμερα το απόγευμα. Η Ευρώπη μεταβάλλεται μπροστά στα μάτια μας και υπάρχει ευξημένο επίπεδο συζήτησης ποια τροπή παίρνει, παίρνουν αυτές οι αλλαγές. Μερικοί αμφισβητούν ακόμα και την επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός χώρος. Χωρίς καμιά αμφιβολία, η ευρωπαϊκή διαδικασία οδήγησε σε μεγάλη επιτυχία ως προς τους βασικούς λόγους για ε, τους οποίους δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πρώτο λόγο, δηλαδή την προώθηση της ειρήνης και σταθερότητας του ευρωπαϊκού χώρου. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιτυχίας δεν μπορεί κανείς πλέον να φανταστεί μια χώρα στην ευρωπαϊκή επικράτεια που να είναι κάπως εκτός. Μου ίσως μήπως φαίνεται αναχρονιστική αυτή η ιδέα λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι τώρα. Αλλά πρόκειται για ε, βεβαίως ένα σημείο στο οποίο πρέπει να φτάσουμε στο τμήμα της Ευρώπης στο οποίο ανήκω στα, στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, στα δυτικά Βαλκάνια. Η συνέχιση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στη δική μας την περιοχή είναι ε, πρώτα απ' όλα ένα μακρόπνο όνειρο ειρήνης, ευημερίας, διαρκούς ειρήνης, σταθερότητας στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι το μόνο πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή η διαδικασία μπορεί να προωθηθεί είναι το πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και προσχώρησης. Αυτή η διαδικασία ελπίζω να συνεχιστεί για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, διότι πρώτα απ' όλα πρόκειται για τον εξευρωπαϊσμό για την υιοθέτηση νόμων και κανονισμών και προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ε, το κεκτημένο, το ευρωπαϊκό και τα κριτήρια της Κοπενχάγης που θα πρέπει να υιοθετηθούν από όλους. Αυτό που είμαι προετοιμασμένος να πω εδώ είναι ότι δεν είναι τόσο το τελικό καθεστώς σε αυτό το στάδιο που έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι η ικανότητα συνέχισης μεταρρυθμίσεων. Ξέρω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, εάν ήρθε η στιγμή για νέα μέλη, αν μπορεί να γίνει διεύρυνση ή όχι, δεν ξέρω σε, αν σε πολλά επίπεδα, σε ποια επίπεδα αυτό θα καταστεί δυνατό και εφικτό, αλλά θα ήθελα να επισμάνω ότι όταν πρόκειται για την ε, Δυτικά Βαλκάνια εκτός από την Κροατία, ε, οι αποφάσεις αυτές δεν είναι για να γίνουμε μέλη, να προσχωρήσουμε ως μέλη σε αυτό το στάδιο βεβαίως. Δεν βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Και νομίζω ότι συνεχιζόμενος εξευρωπαϊσμός της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων είναι νομίζω προς όφελος και των Σέρβων πολιτών αλλά επίσης και προς όφελος όλου του ευρωπαϊκού χώρου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να, να μιλήσω για την σημαντική απόφαση ε, που θα ληφθεί στις 9 Δεκεμβρίου που θα είναι μια ημερομηνία πολύ σημαντική για τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα είναι η ημερομηνία όπου η ε, Κροατία θα υπογράψει τη συνθήκη προσχώρησης. Και παρόλες τις ε, δυσκολίες στον ευρωπαϊκό χώρο, παρόλες τις κρίσεις που πλήττουν την Ευρώπη, Δεκεμβρίου θα, θα έχουμε καλές ειδήσει ε, για τα Δυτικά Βαλκάνια, διότι η Κροατία θα υπογράψει τη συνθήκη προσχώρησης. αλλά νομίζω εξίσου σημαντικό για το θέμα αυτό, όπως και για το θέμα της υπογραφής, είναι το σήμα, το μήνυμα που θα σταλεί από τις Βρυξέλλες σε σχέση με το τι συμβαίνει μετά. Μετά την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί αναλυτές πολλοί άνθρωποι που, που έρχονται από διάφορες προελεύσεις που λένε που πρέπει ε, να υπάρξει μια διακοπή, ένας χρόνος ε, σκέψης, εξέτασης, προβληματισμού, ε, προτού προχωρήστε. η 9η Δεκεμβρίου είναι γεμάτη συμβολισμούς από πολλές απόψεις, ακόμη και από την άποψη της συνέχισης της διαδικασίας διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Στους τελευταίους 24 μήνες στη Σερβία είχαμε 24 μήνες εξαιρετικής πρόοδου θα έλεγα. Υπήρξαν σοβαρές μεταρρυθμίσεις και η, Ευ... η γνωμοδότηση 12 Οκτωβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε την πρόοδο αυτή των 24 τελευταίων μηνών, όπου έλαβαν σημαντικές, χώρα, σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας. Ως προς τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι εξόφθαλμα, κυρίως ε, λόγω της ε, τελευταίας κρίσης στον ευρωπαϊκό χώρο, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Σερβία έχει μειώσει σε 45% τον λόγο χρέους προς το ΑΕΠ. Είμαστε η μόνη χώρα μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ που αναβαθμίστηκε ως προς τον κίνδυνο των επενδύσεων από την αρχή της κρίσης και από τις λίγες χώρες στον κόσμο που αναβαθμίστηκαν όσον αφορά την ε, πιστοληπτική ικανότητα. Και αυτό ήταν από την αρχή της κρίσης. Αυτό έγινε μετά την αρχή της κρίσης. Είμαστε λοιπόν υγιείς από την άποψη αυτή και δεν ήταν εύκολο να αναλυφθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις με τις συνθήκες που επικρατούν στον ευρωπαϊκό χώρο. Όσον αφορά την, το δικαστήριο της Χάγης, εδώ είναι ένα θέμα του παρελθόντος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πια τέτοιο πρόβλημα η σερβική κυβέρνηση έχει εργαστεί σκληρά για να συνεργαστεί με το δικαστήριο της Χάγης και ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ε, δεν υπάρχουν πλέον, ε, πλέον νέοι κατηγορούμενοι. Σχετικά με την περιφερειακή συνεργασία είμαι, μπορώ να πω ότι οι σχέσεις ε, στα Βαλκάνια δεν υπήρξαν καλύτερα από την αρχή του, του πολέμου για την διαδοχή της Ιουγκοσλαβίας το 1981 και αυτό έχει να κάνει με την σκληρή προσπάθεια των ηγετών της χώρας αυτής και των χωρών αυτών. Η Σερβία έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία συμφιλίωσης. Και ακόμη, όταν πρόκειται για τα πιο λεπτά θέματα του Κωσοφοπεδίου. Νομίζω ότι συζητήσατε το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, πολύ λεπτό ε, για τα εμπλεκόμενα μέρη. Νομίζω ότι ακόμη και σε αυτό το τομέα έχει πραγματοποιηθεί σοβαρή πρόοδος από την αρχή ε, του διαλόγου μεταξύ Βελιγραδίου και Πριστίνας υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διάλογος αυτός άρχισε ε, μεταξύ των 27 χωρών και της Σερβίας και της, ε, του κοινού ψηφίσματος που υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Άρχισε ο διάλογος και για πρώτη φορά στην ιστορία άμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δύο μέρη άρχισαν να αποφέρουν καρπούς. Αυτό πολύ συχνά υποτιμάται και θα ήθελα να τονίσω την σημασία της δέσμευσής μας σε αυτό το διάλογο και όλων των εμπλεκομένων μερών. Νομίζω ότι ενέχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι ο διάλογος αυτό συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ε, μερικές πολύ σοβαρές διαφορές και απόψεις μεταξύ των μερών. Δεν θέλω όμως ε, να ξοδέψω πολύ χρόνο μιλώντας. Είναι σημαντική απόφαση ως προς τα Δυτικά Βαλκάνια η απόφαση αυτή της 9ης Δεκεμβρίου. Ελπίζω ότι θα έχουμε καλές ειδήσει και για την Σερβία σε αυτή τη συνάντηση. Εάν δεν συμβεί αυτό, δεν θα είναι το τέλος του κόσμου για κανέναν. Η Σερβία μιλάω εξ ονόματος αυτής της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αυτή θα παραμείνει δεσμευμένη στο ευρωπαϊκό μέλλον και νομίζουμε ότι το, η ευρωπαϊκή διαδικασία είναι προς συμφέρον των πολιτών μας και προς όφελος της γεωγραφίας της εθνικής, της τοπικής, της περιφερειακής, της υπηρετικής. Και αυτό έχει να κάνει με την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής προσπάθειας της προσπάθειας που αποβλέπει ε, στο ευρωπαϊκό μέλλον των Βαλκανιών των κοινών μας προσπαθειών, προσπαθειών της Σερβίας, των γειτόνων μας, των εταίρων μας. Νομίζω ότι είχαμε 24 μήνες εξαιρετικούς στο παρελθόν μας και ελπίζω ότι θα έχουμε και άλλους 24 μήνες ε, στο μέλλον που θα είναι εξαιρετικοί αν βρούμε ε, το θάρρος και τη δύναμη να συνεργαστούμε και να ε, υπερνικώντας τις δυσκολίες να προοδεύσουμε προς όφελος των κοινών μας αξιών. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ε, δεν θα έχουμε πολύ χρόνο δυστυχώς στη διάθεσή μας για προφανείς λόγους. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας με τη χώρα σας, ο κύριος Κουκάνα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Σας καλωσορίζω κύριε Υπουργέ Γέρεμιτς. Καλωσορίζω την πρέσβη της Σερβίας. Είναι πολύ σημαντική η στιγμή και για τη Σερβία και για τα υπόλοιπα Βαλκάνια και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο χρόνος ανάμεσα στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου νομίζω ότι έχει σημασία. Πάρα πολλά θέματα επηρεάζουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και προς τη θετική κατεύθυνση. Ελπίζω ότι τα συμπεράσματα αυτά θα είναι πάρα πολύ καθοριστικά για τη Σερβία και τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Κατανοώ την περιπλοκότητα της πολιτικής κατάστασης στη χώρα σας, οι εκλογές τον επόμενο χρόνο, ένταση στον βορρά του Κωσυφοπεδίου, προεκλογική εκστρατεία, όλα αυτά είναι θέματα, αλλά θα θέλαμε πράγματι να δούμε μια Σερβία η οποία να ακολουθεί την ευρωπαϊκή πορεία και όλοι θα θέλαμε να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ξέρω ότι δεν είναι ε, εύκολο να προχωρήσει κανείς με επιτυχία στις εκλογές προωθώντας ε, φιλοευρωπαϊκά συνθήματα σε αυτή τη φάση. Είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή που βιώνουμε τώρα και είναι κάτι το οποίο θα θέσει θα έλεγα σε δοκιμασία την πολιτική σας οριμότητα και ελπίζω να μπορέσετε να προχωρήσετε. Θα ήθελα μία ερώτηση να θέσω. Όλοι είδαμε την έκθεση. Πώς αξιολογείτε την επίδοση της κυβέρνησής σας στα πλαίσια της διαδικασίας εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών κριτηρίων. Πώς το βλέπετε εσείς όμως από τη δική σας πλευρά. Ευχαριστώ. Πράγματι λίγα δευτερόλεπτα καθυστερήσανε. Ο κύριος Κασίν, εισηγητής για τη Σερβία. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ, κύριε Πρέσβη. Θέλω να σας συγχαρώ για όλα αυτά τα οποία πέτυχε η χώρα σας στους τελευταίους μήνες και να σας ε, πληροφορήσω ότι θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε την πρόοδο στη χώρα σας. Γι' αυτό τον Ιανουάριο έχουμε την πρώτη ανάγνωση της έκθεσης πρόοδου της Σερβίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα τελειώσει αυτή η διαδικασία στο τέλος Μαρτίου. Ε, τους επόμενους τρεις μήνες λοιπόν θα έχουμε πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τη Σερβία. Θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε πλήρωστη στη χώρα σας. Εγώ ελπίζω εκ καρδίας ότι μετά από την 9η Δεκεμβρίου θα έχετε όχι μονάχα γείτονε που θα είναι πια de facto μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ρουμανία και Κροατία βέβαια, και δύο υποψήφιες χώρες όμως, και ελπίζω θα είστε κι εσείς μια υποψήφια χώρα, στην περιοχή των Βαλκανίων. Ελπίζω ότι το Μαυροβούνιο θα πάρει τη σκητάλη από την Κροατία και θα ξεκινήσει διαπραγματεύσει. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Περιοχή σας. Έχω ένα ερώτημα όμως για σας επίσης, γιατί συζητούσα πριν από μία ώρα με τον Σλόμπαντον Πέτροβιτς, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Κωσικοπεδίου, για την εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν συναυθεί μέχρι στιγμής. Όπως ξέρω πριν από λίγες μέρες η νομική σας υπηρεσία προετοίμασε μια, την θέση του Υπουργείου σας σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών και φαίνεται ότι έχετε σημαντικές επιφυλάξεις για τη δυνατότητα εφαρμογής αυτών των συμφωνιών γιατί δεδομένου ότι όλοι περιμέναν ότι εσείς θα εφαρμόσετε όλες αυτές τις συμφωνίες θα ήταν πολύ χρήσιμο για μας να ακούσουμε από τη δική σας πλευρά μία εξήγηση για το θέμα αυτό. Είσαστε τμήμα της λύσης ή τμήμα του προβλήματος. Είναι εφικτό αυτό να υλοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες ή όχι. Εμείς είμαστε εδώ ως υποστηρικτές της Σερβίας και θέλουμε σε 9 Δεκεμβρίου να γιορτάσουμε μια επιτυχία. Αλλά πέστε μας, θα είναι πραγματικότητα ή θα είναι άπια στο όνειρο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπροκ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπατε και μπορείτε να είστε σίγουρος ότι και η δική μου πολιτική ομάδα υποστηρίζει την τήρηση των υποσχέσεων της Θεσσαλονίκης του 2003. Όλα αυτά έχουν σαν στόχο να εξασφαλίσουν και τη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων. Και αυτό φυσικά είναι και προ το συμφέρον της Ευρωπαϊκή Ένωσης να υπάρξει εξέλιξη προς την κατεύθυνση της σταθερότητα στην περιοχή. Και γι' αυτό ενδιαφερόμαστε και για, τι μεταρρύθμιση, τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν στις χώρες αυτές, που έτσι κι αλλιώς έχουν νόημα, ακόμα και αν δεν, θα είχαν νόημα ακόμα και αν δεν υπήρχε προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να γίνουν προς όφελος των πολιτών των χωρών αυτών. Η εξασφάλιση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της καταπολόμησης, της διαφθοράς, η οικονομική ανάπτυξη, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον πληθυσμό των χωρών αυτών και όχι μοναχά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η ευρωπαϊκή προοπτική μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη στο πλαίσιο αυτό των μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι οι εξελίξεις που στρέφονται κατά των εθνικισμών και είναι υπέρ της ειρηνικής λύσης των προβλημάτων, προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο, παραδείγματος χάρη, είναι ένα θετικό βήμα και έφεραν όλα αυτά τη Σερβία πολύ κοντύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι και μετά την προκήρυξη της χώρας ως υποψήφιας χώρας υπάρχουν πολλά κόμματα τα πρέπει να επιτευχθούν. Αλλά δεν είναι πια απομεμακρυσμένος στόχος η ένταξη της Σερβίας. Είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί ο ενδιάμεσος στόχος του καθεστώτος υποψήφιας χώρας και σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ελέγχθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές, θα ήθελα να σας ρωτήσω και σε σχέση ιδιαίτερα με το κοσφοπέδιο, πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην περιοχή σας και ιδίως τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την ελίπουσα ικανότητα της κυβέρνησης στη Βοσνία Σεγοβίνη να δημιουργήσει μια κυβέρνηση. Είναι έτοιμη να ξεπεράσει το Βέλγιο η Βοσνία Ζεγοβίνη σε ό,τι αφορά το χρόνο δημιουργίας κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιγγενίν. Ένα λεπτό, μισή λεπτό μόνο. παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ Γέρεμιτς και εξ ονόματος των Σοσιαλδημοκρατών στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που βρήκατε χρόνο για να συζητήσετε μαζί μας. Περιμένουμε και εμείς όπως και εσείς τις αποφάσεις του Συμβουλίου για τον επόμενο μήνα. Ако си спомним откъде тръгнаха процесите и къде са днес, смятам, че усилията и на Όταν δούμε τι εξελίξεις έχουν υπάρξει και όταν δούμε το πώς έχουν πράγματι προχωρήσει τα πράγματα, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε μια τεράστια προσπάθεια την οποία έχετε κάνει και γι' αυτό ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας έδωσε την ιδιότητα της υποψηφίας χώρας. Ξέρω ότι η περίοδος στην οποία βιώνετε δεν είναι εύκολη. Ένα από τα πιο βασικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να υποστηρίξει την κυβέρνησή σας έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί σωστά τις προσδοκίες των λαών της Σερβίας. Οι πολίτες αυτοί πρέπει να νιώσουν την ελπίδα για ένα ευρωπαϊκό μέλλον και πράγματι αν σας δοθεί ο τίτλος της υποψηφίας χώρας, αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα, θα είναι ένα κίνητρο για τη Σερβία, θα είναι ένα σημαντικό εν πάση περιπτώσει βήμα, ξαναλέω, στην πορεία για την ένταξη. Δεν θα ήθελα να συνεχίσω μια τέτοιου είδους ανάλυση της κατάστασης. Αυτό που θα συμβεί στη χώρα σας είναι σημαντικό και για όλη την περιοχή. Υπάρχουν βέβαια ορισμένε χώρες οι οποίες αμφισβητούν τις προσπάθειες τις οποίες κάνετε. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Γνωρίζετε τα μηνύματα τα οποία στέλνουν, σας στέλνουν οι χώρες αυτές τι θα κάνει η κυβέρνησή σας μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου έτσι ώστε να πείσετε αυτές τις χώρες οι οποίες είναι, έχουν αμφιβολίες να στηρίξουν την υποψηφιότητά σας. Ευχαριστώ η κυρία Λούνατσεκ. Εσείς θα μπορέσετε να χωρέσετε στο 1,5 λεπτό. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τον Υπουργό της Σερβίας ε, και τον Πρέσβη και συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι 9η Δεκεμβρίου θα είναι μια, σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Σερβία αλλά και για τα Βαλκάνια, την Κροατία διότι η Κροατία θα υπογράψει τη Συμφωνία Ένταξης και ε, ελπίζω η Σερβία και το Μαυροβούνιο ε, να πάρουν το καθεστώς ε, του υποψηφίου χώρας και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Χαίρομαι που ο Επίτροπος Φούλε στην έκθεση προόδου είπε ότι συνιστά το καθεστώς αυτό για τη Σερβία, αλλά πρέπει να γίνει πρόοδος στον διάλογο με το κοσυφοπέδιο. Και εσείς υπήρξατε σαφείς και χαιρετήσατε την όλη διαδικασία διαλόγου, κύριε και είπατε ότι ε, η Σερβία συμφώνησε πριν από ένα χρόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Νέα Υόρκη. Ε, το θετικό είναι ότι είναι θετικό το βήμα αυτό. Το πρόβλημα που έχω, ότι είναι, ξέρω βεβαίως ότι άρχισαν οι συναντήσεις, αλλά η Συμφωνία των Αρχών Ιουλίου δεν έχει εφαρμοστεί από την Σερβία. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορείτε να εξηγείτε, εξηγήσετε ότι ο διαπραγματευτής κ. Σοφάνοβιτς μπλόκαρε την συνάντηση των διαλόγου, ε, μην, μη δεχόμενος τις σφραγίδες ε, των ε, τελωνίων που δεν γίνανε δεκτές από την ΟΝΜΙΚ και στάλησαν στην δική σας κυβέρνηση. Αυτό θα πρέπει να το έχει κάνει η Σερβία εδώ και αρκετό χρόνο. Ε, και πάρα πολλά από αυτά τα θέματα δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Θα σας ζητούσα να μα πείτε πώ ε, όλα αυτά τα πράγματα θα εφαρμοστούν από την Σερβία τις επόμενες μέρες, διότι χωρίς αυτά Νομίζω ότι θα είναι προβληματική η κατάσταση της Σερβίας και τα κράτη-μέλη ίσως έχουν επιφυλάξεις για να δώσουν το καθεστώς υποψηφίας χώρας στην Σερβία. Χρειάζονται εφαρμογές, υλοποίησει και όχι μόνο συμφωνίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να καλωσορίσω εδώ τον Υπουργό Γέρεμιτς. Συγχαίρω τη χώρα σας ε, για την οικονομική της ανάπτυξη, την βελτίωση της διακυβέρνησης, παρόλο που υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με την διαφάνεια των αποκρατικοποίησεων και το γεγονός ότι μπορέσατε να αναπτυχθείτε ε, παρά τους αντίθετους ανέμους που πνέουν διεθνώς λόγω της παγκόσμιας κρίσης και κυρίως την κρίση εδώ στην Ευρωζώνη. Η ομάδα μου υποστηρίζει το, το να γίνεται υποψήφια χώρα μαζί με την Μακεδονία και το Μαυροβούνιο και όλες αυτές οι χώρες θα πρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις σύντομα. Βεβαίως υπάρχουν τα εμπόδια που γνωρίζουμε σχετικά με την Μακεδονία. Η Κροατία έχει προχωρήσει αλλά βεβαίως αντιμετωπίζουμε ε, μια κόπωση ως προς την ε, διεύρυνση. Ανέφερα την ε, κρίση της Ευρωζώνης που είναι το θέμα που απασχολεί τους ηγέτες μας εδώ και βεβαίως και η διαδικασία μεταρρύθμισης στις χώρες σας προτού δεχθούμε μια άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα Δυτικά Βαλκάνια. Το θέμα του διαλόγου Βελιγραδίου Πριστίνας, στο οποίο αναφέρθηκαν Αναφέρθηκε και η Βαρόνη Άστον. Τι συγκεκριμένα αποτελέσματα περιμένετε από αυτές τι συνομιλίε. Μέχρι τώρα είδα πάρα πολύ λίγα πράγματα και συμμερίζεστε την προσωπική μου άποψη ότι η διεθνή ε, κοινότητα δεν θα έχει πια υπομονή ε, ε, χρηματοδοτώντας την παρουσία στο κοσυφοπέδιο και ότι αργά ή γρήγορα ε, θα ε, πρέπει να γίνει κάποια ανταλλαγή για την ειρήνη και να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σεβερίν για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Με την πρόοδο της Σερβίας για την επίτευξη των δικών της προσδοκιών και των δικών μας προσδοκιών. Αυτή η πρόοδος φυσικά εξαρτάται από τις προσπάθειες των Σέρβων. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο περισσότερο σε σχέση με την, με εικόνα που έχει η κοινωνία της Σερβίας εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θεωρούν ότι τα ανοίγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Σερβία έχουν συνεχτικό χαρακτήρα και αν αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Σερβία για να υλοποιήσει τις, υποσιο... τις υποσχέσεις της. Και θεωρώ ότι αυτό το ερώτημα θα πρέπει να τύχει και κάποιες απάντησεις και στο φως της πρόσφατης παράδοσης του στρατηγού Μλάντιτς που ήταν ένα σημαντικό βήμα. Μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σέβεριν η κυρία Κόπα, η οποία είναι σκιώδης εισηγήτρια για τη Σερβία. Παρακαλώ ένα λεπτό μονάχα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να χαιρετήσω τον Υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας και φυσικά να συγχαρώ τη Σερβία για την πρόοδο που επέτυχε τον τελευταίο χρόνο σε επίπεδο δημοκρατικοποίησης, σε επίπεδο συμφιλίωσης και σε επίπεδο πλήρους συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το ερώτημα μου αφορά και πάλι το κοσφοπέδιο. Χαιρόμαστε που τώρα ξανά άρχισε ο διάλογος. Όλοι ελπίζουμε θα υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε από τα μέσα ενημέρωσης και από άλλα, άλλες πηγές είναι κάπως αντιφατικές πληροφορίες. Ποια είναι η δική σας ε, ανάγνωση των γεγονότων και ποιο είναι το σχέδιό σας για το μέλλον. Μπορούμε να περιμένουμε και να προστοκούμε θετικές εξελίξεις μέσω από τη διαδικασία διαλόγου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Κόπα. Κύριος Κόβατσακ, για ένα λεπτό μονάχα. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν με βλέπετε, είμαι εδώ. Η πλειοψηφία αυτού του κοινοβουλίου, λέει ο κ. υποστηρίζει τις ε, προσπάθειες που κάνετε για να πορευτείτε προς τη δημοκρατία στη Σερβία και ελπίζουμε ότι ήδη από το 1912 θα συνεχίσετε την προσπάθεια αυτή για μια ακόμα πιο φιλοευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας. Ελπίζω να μην μείνετε απλά στο καθεστώς της, ε, του, της υποψήφιας χώρας, αλλά κάποια στιγμή να γίνετε και μέλος της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να αναφερθώ εδώ και στις εμπειρίες τις οποίες έχει βιώσει η δική μου χώρα μια κομμουνιστική χώρα με ισχυρές ε, αστυνομικές δυνάμεις και μυστικές υπηρεσίες. Ε, τι γίνεται με το παρελθόν στη Σεβία. πώς αντιμετωπίζετε τα προβλήματα. υπάρχουν ε, σχέσεις ανάμεσα ας πούμε στην διπλωματική υπηρεσία της Σερβίας και στην παλαιά δομή της ε, ε, ε, κατασκοπίας και τα λοιπά. Ξέρω ότι από πλευράς της ΦΥΡΟΜ έχει ζητηθεί από την Σερβία να της δώσουν κάποια αρχεία τα οποία φυλάσσονται στο Βελιγράδι και είναι σχετικά με την σημερινή ΦΥΡΟΜ και που αφορούν την δράση των πολιτών της χώρας αυτής εκείνη την εποχή. Και επίσης θα ήθελα να αναλύσετε λίγο και ε, για τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει για την ανάκτηση της, ε, ανάκτηση της ιδιότητας του Σέρβου πολίτη από τους κατοίκους Κοσφοπεδίου. Παλέσκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. στην ε, παρέμβασή σας αναφερθήκατε στο γεγονός ότι το κοσφοπέδιο είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα. Θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Όπως ξέρετε, η Ρωσία θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος παραλληλισμός μεταξύ της κατάστασης του κοσφοπεδίου και της καταστάσεως στην Βόρεια Οσετία ή Απχαζία. Ποια είναι η δική σας άποψη λοιπόν για την Απχαζία και τη Βόρεια Οσετία και το καθεστώς τους. και τι είδους επικοινωνία υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Βελγραδίου και Μόσχας για τα θέματα αυτά. Ο κύριος Στόκας. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον ε, κύριο Υπουργό. Εμείς έχουμε συναντηθεί ήδη με την ε, κυρία Πρέσβη που βρίσκεται στο πλευρό σας και έχουμε μιλήσει για αυτή την ποινική διαδικασία που έχει χαρακτήρα διακριτικό. Και έχουμε πάρα πολλές αμφιβολίες και ανησυχίες αυτή τη στιγμή για αυτή την, την διαδικασία συλλογικής, συλλογικών κυρώσεων η οποία ε, κινδυνεύει να επαναφέρθει. Ποιες είναι οι προοπτικές αυτή τη στιγμή. Έχετε καταφέρει να επιλύσετε τα προβλήματα που υπήρξαν στο παρελθόν με την Ουγγρική μειονότητα. Στο εδαφό σα. είχαμε τα ίδια προβλήματα στην, ε, στη Ρουμανία και τα βλέπουμε τώρα στην ε, Σερβία. Αυτοί οι οποίοι ζουν λοιπόν στην περιοχή του Τιμοκλάκ είναι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι οι βλάχοι οι οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Οι τελευταίες απογραφές κατέδειξαν ποια είναι και η κατάσταση του πληθυσμού ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Όρμπαν, έχει τονίσει τη σημασία του να μην μείνει σαν μια μαύρη τρύπα το κομμάτι των Δυτικών Βαλκανίων, τελευταίος ομιλητής κυρία Μποσκούρτ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εκπρόσωπο της Σερβίας γιατί η χώρα του έχει κάνει σημαντικά βήματα. Έχω δύο ερωτήματα τώρα για τα κριτήρια της Κοπεχάης και την δυνατότητα να γίνει μέλος της Σερβία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γεγονός ότι οι χώρες οι οποίες έχουν συγκρούσεις ανοιχτές έχουν ένα πρόβλημα και αυτό είναι και το ερώτημα το οποίο θα σας θέσω για το κοσφοπέδιο και είχα ζητήσει στο παρελθόν για την περιοχή του Σάντζα και είπατε ότι και εκεί η κατάσταση είναι δύσκολη. Πώς λοιπόν μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς αυτά τα προβλήματα αυτό είναι απαραίτητο και για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το, θέμα, το άλλο θέμα είναι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι όλο και περισσότερε περιπτώσει οι οποίε προέρχονται από τη Σερβία και έρχονται ενώπιον των διεθνών δικαστηρίων. Μπορείτε να μα εξηγήσετε γιατί υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα. Θα αφήσουμε τον απαραίτητο χρόνο. Δεν είναι επαρκής βέβαια δεν είναι ο χρόνος που χρειαζόστε, αλλά θα σας δώσουμε λοιπόν το χρόνο που χρειάζεται για να μπορέσετε να απαντήσετε σε αυτά τα πολυπληθή ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να απαντήσω τα περισσότερα από αυτά τα ερωτήματα. Είναι τόσα πολλά αυτά τα ερωτήματα που θα ήθελα να ξεκινήσω απαντώντας τα πιο εύκολα ερωτήματα. Το πιο εύκολο ερώτημα είναι αυτό του κυρίου Κούκαν. Φυσικά δεν μπορώ παρά να είμαι υποκειμενικός γιατί είμαι μέλος της σερβικής κυβέρνησης, της τρέχουσας σερβικής κυβέρνησης. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Η σωστή αξιολόγηση πρέπει να γίνει από κάποιους άλλους. Είναι πιο αντικειμενική άμα γίνεται από κάποιους άλλους από εμά, αλλά νομίζω ότι ένα καλό ε, σημείο φαίνεται στην ε, γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέει πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Σερβία έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της βάσει της Συμφωνίας Σταθεροποίησης. Δεν είναι εύκολη εποχή για να μπορείς κανείς να τηρήσει τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι απαιτείται και αν μας δοθεί η ευκαιρία ο λαός της Σερβίας θα συνεχίσει και τον επόμενο χρόνο να προχωρήσει το δρόμο αυτής της διαδικασίας μεταρρύθμισης. Για τα θέματα της συμφιλίωσης, νομίζω ότι έχουν γίνει κάποια ε, βήματα χωρίς προηγούμενο τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την συμφιλίωση. Και θα παραμείνουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και τις πεπιθήσεις μας και στους στρατηγικούς μας στόχους. Αν αυτό θα μας φέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλα. Ποια θα είναι η σειρά αλλά το να ευρωπαϊκοποιήσουμε τη Σερβία, να την ευθυγραμμίσουμε σε νομοθετικό επίπεδο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι μόνο για τη Σερβία, αλλά όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα ανεξάρτητα από τις πολιτικές δυσκολίες που μπορεί να υφίστανται αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσω να απαντήσω δύο ή τρία ερωτήματα που είναι παρόμοια. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κατσίν για την προσήλωσή του στο ευρωπαϊκό μέλλον της Σερβίας, όπως και αυτός εμείς πάντα κάνουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια να είμαστε τμήμα της λύσης και όχι τμήμα του προβλήματος. η συμφωνία που έγινε και οι συμφωνίες που θα συναυθούν στο μέλλον στο διάλογο μεταξύ του Βελιγραδίου και της Πρίστινα θα πρέπει να συνάδουν με κανόνες, με νομοθεσία, με το Σύνταγμα της Σερβίας και με τους νόμους της Σερβίας. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη γνωμοδότησή της ότι το Σύνταγμα και το νομοθετικό πλαίσιο της Σερβίας ευθυγραμμίζεται σε γενικό βαθμό με τις απαιτήσει Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ανεπτυγμένο το νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει να σεβαστούμε λοιπόν αυτούς τους νόμους και αυτό το πλαίσιο. Μία από τις βασικές ευρωπαϊκές αρχές είναι ο σεβασμός των κανόνων. Αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε σε οποιαδήποτε πτυχή των προσπαθειών μας είναι να εξασφαλίσουμε το σεβασμό του νόμου. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας υπόψη μας την διαπεπραγματευμένη λύση αυτής της πάρα πολύ δύσκολης κατάστασης. Ο διάλογος αυτός έχει λοιπόν την ευκαιρία, τη δυνατότητα να αποβεί επιτυχής. Μέχρι στιγμής ήταν επιτυχής σε πολλούς τομείς. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα τα οποία πρέπει ακόμα να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν μέσα στο διάλογο αυτό. Πολλά εκρεμή θέματα θα ήθελα να αντιμετωπιστούν προτού ληφθεί μια απόφαση από τις αρχές της Πρίστινα για μια μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας γιατί θα ήταν καλύτερη κατάσταση τώρα αλλά τα πράγματα είναι όσοι έχουν τώρα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε με την καλή την πίστη με τον καλύτερο τρόπο όλα αυτά τα ανοιχτά θέματα. Και θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι ο λόγος για τον οποίο μπορέσαμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε 28 χώρες, έξι από τις οποίες έχουν μία άποψη για την ανεξαρτησία του πεδίου, της λεγόμενης μάλλον δημοκρατίας του πεδίου, και 22 χώρες έχουν μία διαφορετική άποψη, ο λόγος για τον οποίο μπορέσαμε να ξεκινήσουμε ένα διάλογο είναι γιατί θεωρούσαμε πρέπει να βρεθούν λύσεις στα ανοιχτά προβλήματα για να μπορέσουν να βρουν κάποια ομαλότητα οι πολίτες της περιοχής. Δεν είναι μια απλή άσκηση για να αποδειχθεί ότι το κοσφοπέδιο είναι ανεξάρτητο κράτος. Ούτε είναι μια άσκηση απόδειξης του ότι το κοσφοπέδιο είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της Σερβίας βάσει των νόμων και των κανόνων μας. Αν μπορέσουμε να κάνουμε πρόοδο στην επίλυση αυτού του προβλήματο για να βρούμε κοινό έδαφο μεταξύ των μερών, ίσως θα μπορέσουμε να είμαστε επιτυχείς. Και πάλι, δεν θέλουμε να δείξουμε ότι μια πλευρά έχει δίκιο ή η άλλη πλευρά έχει δίκιο. Είναι μια προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει κάποια ομαλότητα στην καθημερινή ζωή των πολιτών που ζουν εκεί, παρά τις πολιτικές διαφωνίες, οι οποίες είναι θεμητές αυτές οι διαφωνίες, και οι οποίες αντανακλούν τη δημοκρατική θέληση των κοινωνιών μας. Για να απαντήσω το ερώτημα του κύριου Μπροκ και ελπίζω κάποιος να το διαβιβάσει. Η Σερβία συμμετέχει ενεργά σε περιφερειακές ενέργειες και εγχειρήματα και έχει παίξει σημαντικό ρόλο και αυτό το λέει η γνωμοδότηση Κομισιόν προεδρεύει των περισσότερων διαδικασιών που γίνονται μέσα στην ε, περιοχή των Βαλκανίων, διάφορες πρωτοβουλίες ευρωπαϊκού χαρακτήρα και μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει διαμαρτυρηθεί για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε ασκήσει την προεδρία αυτών των φορέων ανεξάρτητα παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο έχουμε κρατήσει την Προεδρία σε αυτό τον πολύπλοκο χώρο χωρίς κανείς να δυσαρεστηθεί δίνει μια καλή αίσθηση του πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουμε τις υπευθυνότητές μας και τον περιφερειακό μας ρόλο και πώς θα ταινίσουμε το μέλλον του τμήματος αυτού των Βαλκανίων. Για τη Βοσνία Ζεχοβίνη η θέση μας είναι πάρα πολύ σαφής. Εμείς σεβόμαστε την κυριαρχία και την εδαφική ακαιρεότητα του κράτους αυτού όπως και οποιοδήποτε άλλου κράτους που είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι και μια απάντηση για το ερώτημα σε σχέση με την Αυχαζία και την ε, Βόρεια Οσετία. Σεβόμαστε την τελική πράξη του Ελσίνσκι, και την διαδικασία που ακολούθησε, όλα τα κράτη έχουν το δικαίωμα σεβασμού στην κυριαρχία τους και την εδαφική τους ακεραιότητα χωρίς καμία εξαίρεση. Δεν μιλάμε ούτε για... Όλα αυτά εφαρμόζονται και στη Σερβία και στη Βοσνία και σε όλα τα κράτη του κόσμου. Προσπαθώντας να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Λούνετσεκ για την εφαρμογή, την υλοποίηση ε, πίσω μας είχαμε μερικούς πολύ δύσκολους μήνες. Και ξέρετε, αν έχετε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που συνεχίζεται, τότε περιμένετε ότι τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό το χώρο ε, θα είναι εμπόδια στην, ε, στην διαδικασία διαπραγμάτευση. Όταν συνεχίζεται και προσκρούει σε εμπόδια αυτή η διαδικασία, τι γίνεται. Αυτό που συνέβη στις 25 Ιουλίου ήταν μια μαζική κίνηση των, του Ρόσολ, των μονάδων των ειδικών του κοσυφοπεδίου στο έδαφος τους, αυτό χωρίς προειδοποίηση ούτε στην Ιούλεξ, ούτε στην ΚΕΙΦΟΡ, 4 ούτε στους βασικούς διεθνείς πρωταγωνιστές. Και το θέμα είναι, προσπαθεί κανείς να επιλύσει τα θέματα στο διάλογο ή στέλνοντας ε, ένοπλες δυνάμεις. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στο διάλογο, Βεβαίω, δεν είναι σαν να περπατάει κανεί σε ένα πάρκο. Προσπαθούμε να διευθετήσουμε θέματα τα οποία συσσωρεύτηκαν, τα οποία ε, υπάρχουν εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Εάν ένας γύρος του διαλόγου δεν φέρει αποτέλεσμα ε, που να αρέσει σε ένα μέρος, αυτό ε, σημαίνει ότι ο άλλος πρέπει να στείλει στρατά. Έστειλαν τις στρατιωτικές δυνάμεις, αυτό δημιούργησε αναταραχή, δημιουργήθησε σε όλο τον πληθυσμό αυτού του τμήματος της επικράτειας στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο να βγει στους δρόμους και να μπλοκάρει τους δρόμους και τα πάντα. Ξέρετε, 97% των πολιτών αυτού του τμήματος της ε, επικράτειας έχουν ε, πολύ συγκεκριμένες απόψεις για το μέλλον ε, του τμήματος αυτό και αν στέλνονται στρατιωτικές δυνάμεις όταν δεν μας αρέσουν τα αποτελέσματα ενός διαλόγου δεν θα προχωρήσουμε πάρα πολύ. Τον Ιούλιο λοιπόν, τι αυτό που συνέβη ήταν δημιούργησε μια κατάσταση όπου η σταθερότητα υπονομεύτηκε σημαντικά. Αυτή δεν είναι μια ατμόσφαιρα που είναι ε, πρόσφορη ε, προς ε, το, διάλογο και τα αποτελέσματά του. Τα περισσότερη ενέργεια μας και ο χρόνος μας αφιερώθηκαν για να υπερνικήσουμε την κρίση στο Βορρά και που ε, ε, επιδεινώθηκε με την εισβολή της στρατιωτική, που δεν είχε συζητηθεί εκ των προτέρων με κανέναν. Όπως είπα, η υλοποίηση για ορισμένα θέματα έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Τον περισσότερο χρόνο τον αφιερώσαμε για να βελτιώσουμε τις επιπτώσεις της μονομερούς διακήρυξης της Πρίστινα μιλώντας στο διάλογο για το πώς ε, να θα υλοποιήσουμε τα αποτελέσματα. Έχουμε ομάδες ε, υλοποίησης, έχουμε ομάδες εργασίας για την εφαρμογή των συμφωνιών που συνάφθηκαν. Βεβαίως θέλουμε να προχωρήσουμε καλή την πίστη σε αυτήν την διαδικασία διαλόγου με δίκαιο τρόπο σύμφωνα με τις κοινέ αξίες και τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή η δέσμευση για να γίνουν όλα αυτά δεν έχει σχέση με το ευρωπαϊκό μας μέλλον. Αυτά τα χρειαζόμαστε, τα αποτελέσματα για να μπορέσουμε να έχουμε μια ομαλή ζωή, να έχουμε σταθερότητα, ε, να έχουμε την ομαλότητα σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Βεβαίως, η επίλυση αυτού του προβλήματος δεν πρόκειται να επιταχύνει την διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν αφελές εκ μέρους μας να περιμένουμε ότι η επίλυση του προβλήματος του κοσυφοπεδίου θα διεκπαιρεώσει την όλη διαδικασία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, αλλά έχουμε δεσμευθεί να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, όπως επίσης δεσμευθήκαμε ε, να επιλύσουμε το θέμα της συνεργασίας με το δικαστήριο της Χάγης. Ξέραμε ότι η διευθέτηση αυτού του προβλήματος δεν επρόκειτο να μας προωθήσει ε, πιο πέρα στον δρόμο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν απογοητευθήκαμε, το κάναμε για τον εαυτό μας πάρα πολύ πίστεψαν ότι η διευθέτηση του θέματος συνεργασίας με το δικαστήριο της Χάγης θα επιτάχυνε τη διαδικασία ένταξης. Ξέραμε ότι δεν θα την επιτάχυνε, αλλά προωθήσαμε αυτή τη συνεργασία διότι ήμασταν πεπισμένοι ότι η διαδικασία συμφιλίωσης πρέπει να βασίζεται στην εξέβρεση της αλήθειας και αυτοί που έχουν διαπράξει εγκλήματα έπρεπε να πληρώσουν το τίμημα για αυτά τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει στο παρελθόν. Το ίδιο με το κοσυφοπαίδιο. Ξέρουμε ότι δεν θα επιταχύνει την ευρωπαϊκή μας πορεία, αλλά πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα αυτά, διότι κανείς δεν θέλει μια ε, παγωμένη διαμάχη. Και έχουμε δεσμευθεί για το θέμα αυτό να το επιλύσουμε με ειρηνικά και διπλωματικά μέσα, όπως δεσμευθήκαμε και στο παρελθόν. Μιλώ βεβαίως πάντοτε εξ ονόματος αυτής της κυβέρνησης. Κάποιος έθεσε ένα θέμα ε, για το αν θα χάσουμε την υπομονή μας. Δεν μπορούμε να χάσουμε την υπομονή μας, γιατί δεν έχουμε πουθενά αλλού να πάμε. Έχουμε, θα παραμείνουμε δεσμευμένοι ε, για να λύσουμε όλα τα προβλήματα των Δυτικών Βαλκανίων για να εξυπηρετήσουμε την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή αυτή του κόσμου, στην Ήπειρό μας. Σχετικά με την εδαφική αυτή διαίρεση είμαστε κατά της διχοτόμησης ε, των κρατών. Και ε, δεν υποστηρίζουμε την διχοτόμηση σε κανένα μέρος, σε καμιά χώρα του κόσμου. Ούτε καν στην δική μας χώρα, την Σερβία. Γι' αυτό είχαμε, έχουμε αντιτεθεί στην μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας του Κωσυφοπεδίου. προσωπικότητα για τους Σέρβους στο Κωσυφοπέδιο, οι Σέρβοι που ζήτησαν την ρωσική υπηκότητα. Νομίζω ότι αυτή η έκκληση παρεξηγήθηκε. αυτή οι Σέρβοι δεν θέλαν να μεταμναστεύσουν στην Ρωσία, να αλλάξουν τον τόπο διαμονής τους. Αισθάνονται ότι είναι απροστάτευτοι. Αυτή ήταν μια έκκληση για προστασία επειδή και νομίζω ότι είναι σοβαρό το θέμα αυτό, το ότι αισθάνονται απροστάτευτοι και χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να εκθέσω το θέμα αυτό. Δεν αισθάνονται προστατευμένοι στο κοσυφοπέδιο ε, Σέρβοι. Δεν θα κάναν τέτοια έκκληση μεγάλης κλίμακος αν αισθανόντουσαν προστατευμένοι. Και... Σχέδια για το μέλλον. Τα σχέδιά μας για το μέλλον είναι να κάνουμε περισσότερα στο διάλογο για να παραμείνουμε δεσμευμένοι, να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και ανεξάρτητα από το τι ε, μας περιμένει στο μέλλον με τη διαδικασία αυτή την ευρωπαϊκή. Πιστεύουμε ότι η οθέτηση κανόνων και ε, νομοθεσιών που θα μας εναρμονίσει με το κοινοτικό εκτιμένο Είναι κάτι το καλό για αυτή τη χώρα. Θα εξακολουθήσουμε την εναρμόνιση αυτή. Βεβαίως πόσο θα είμαστε αξιότιμοι, αξιόπιστοι ε, και ισχυροί σε αυτή την ε, προσπάθεια. Και νομίζω ότι από την άποψη αυτή έχουμε καλές ειδήσει. Έχουμε μια καλή όθηση που θα δοθεί από την απόφαση της 9ης Δεκεμβρίου. Και η τελευταία ερώτηση στην οποία θα προσπαθήσω να απαντήσω αναφέρεται στο Σαντζάκα, στη χώρα μας, στην νότιο μέρος. Υπάρχει, υπάρχει ριζοσπαστικό Ισλάμ άνοδός του σε αυτό το τμήμα της Σερβίας. Έχουμε ηγέτες θρησκευτικού εξέχοντες σε αυτό το τμήμα της Σερβίας Ε, που ασκούν μια ρητορική πολύ ριζοσπαστική ε, που παρακινεί στην αστάθεια και στο μίσος σε αυτό το τμήμα της χώρας μας. Συνεργαζόμαστε με τους πολίτες, με τις τοπικές αρχές και έχουμε δεσμευθεί να έχουμε αρμονικές σχέσεις με τις διάφορες εθνότητες, τις διάφορες θρησκείες, όλες τις ομάδες στη Σερβία και ελπίζω ότι θα, θα μπορούμε να τηρήσουμε τους νόμους και τις δεσμεύσεις και με τον πληθυσμό μαζί θα μπορούμε να μειώσουμε το περιθώριο δράσης τέτοιων εξτρεμιστών. Υπάρχουν ε, βεβαίως τέτοιοι εξτρεμιστές σε αυτό το τμήμα του κόσμου. Η ερώτηση σχετικά με τους Ρουμάνους, με τους Βλάχους, είχαμε μια επίσκεψη του Βασέσκου στην Σερβία. Συζητήσαμε το θέμα αυτό λεπτομερός και εργαζόμαστε διμερός με τη Ρουμανία για να βεβαιωθούμε ότι το θέμα αυτό θα επιληθεί στο μέλλον. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τη Ρουμανία και με πνεύμα καλής, καλών σχέσεων μεταξύ γειτόνων θα εξακολουθήσουμε να εξετάζουμε το θέμα αυτό. Ε, σεβόμαστε, καταλαβαίνουμε την άποψη της ρουμανικής κυβέρνησης σχετικά με το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας. Ναι, θα πρέπει να σας απαντήσω διαμέσου της πρεσβείας ε, δεν έχω απάντηση να σας δώσω για την επιστροφή αυτών των αρχείων. Ε, θα, φροντίσω να λάβετε την απάντηση. τα θέματα του παρελθόντος, ε, του κομμουνιστικού παρελθόντος στη Σερβία είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Ήμασταν τυχεροί στη χώρα μας που δεν ζήσαμε τέτοια καταπίεση όπως μερικοί άλλοι. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα αυτό. Ένα θέμα που χρήζει σοβαρής ε, αντιμετώπισης ε, και θα βεβαιωθώ να σας δοθεί μια απάντηση. Αλλά ό,τι να σας πω τώρα δεν ε, θα είναι κάτι το όσο βάσιμο θα ήθελα να είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που επιδείξατε για τη χώρα μας. Ξέρω ότι δεν είσαστε το όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα λάβει αποφάσεις την 9η Δεκεμβρίου, αλλά θα εκτιμούσαμε πολύ την κατανόηση και την υποστήριξή σας στο μέτρο του δυνατού για αυτή τη σημαντική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ κύριε Υπουργέ. Η τελευταία σας ευχή είναι κάτι το οποίο σημεριζόμεθα. Ελπίζουμε το Δεκέμβριο να αναγνωριστούν οι προσπάθειά σας. Θα ήθελα να σας πω εκ των προτέρων ότι προβλέψαμε την οργάνωση μιας αντιπροσωπείας στη χώρα σας στις αρχές του επόμενου έτους. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας επισκεφθούμε πλέον επίσημα σαν υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ευχή την οποία κάνουμε και εμείς αφού σας ακούσαμε και αφού αξιολογήσαμε θετικά τις προσπάθειες τις οποίες κάνουν τα όργανα της χώρας σας για να έλθουν πιο κοντά στην Ευρώπη.